Καλησπέρα. Σήμερα δεν έχουμε πάρα πολλά μέλη στην Επιτροπή μας. Ξεκινάμε με το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Σας επενθυμίζω ότι έχει διανεμηθεί αυτή η ημερήσια διάταξη στους συναδέλφους και ως συνήθως τροποποιούμε το σημείο το 9 ε, πήγε για τις 20 Δεκεμβρίου. Οι ίδιοι οι αναφέροντες το ζήτησαν αυτό. Επεσήμαναν για, ότι θα είναι παρόντες. Οι αναφερόμενοι παρουσίασαν την αναφορά που είναι στα σημεία 6, 7, 8, 10 και 11. Στις 5.30 θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Αύριο το πρωί ε, θα γίνει η συζήτηση με τον Επίτροπο Ποτότσνικ που θα έρθει στην Ακρόαση. Ε, δέχτηκε την πρόσκλησή μας και μετά την ακρόαση του Επιτρόπου Ποτότσνικ θα συζητηθούν αναφορές ε, για τις οποίες θα είναι παρόντες οι αναφέροντες είναι στα σημεία 20, 21 και 23 για αυτές τις αναφορές. Αυτές θα συζητηθούν αύριο. Σας λέω ότι αύριο στις 12.30 θα δεχτώ μια αναφορά όσον αφορά την υγεία των ζώων. Σας το επισημαίνω, διότι ίσως να υπάρχουν συνάδελφοι που ενδιαφέρονται θα γίνει η παράδοση εκτός της αιθούσης, θα μπορέσουν λοιπόν να ε, συμμετάσχουν σε αυτή την επίδοση. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε συγκεκριμένη την σε διάταξη, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Πρέπει μετά να εγκρίνουμε το σημείο 2, τα πρακτικά των συνεδριάσεων, της συνδυάσεω της 8 Σεπτεμβρίου και 3 και 4 Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούνται συγκεκριμένα τα πρακτικά. Όσον αφορά τώρα τα άλλα διανεμημένα έγγραφα που έχουν οι συνάδελφοι, έχετε στην κατοχή σας και αντίγραφο μιας αναφοράς της 481 του 2009 που έχει σαν στόχο τη διεύρυνση της βιομηχανικής περιοχής του Βιλιάντο Κόνο στην Φένεα Λακορούνια ζητήθηκε να ξανανοίξει αυτή η αναφορά από τη συνάδελφο Γιονκέρας και η Τουργκάης, ο κύριος Ιτουργκάης ζητάει να παρέμβει. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, είναι μια αναφορά που είχε κλείσει στο παρελθόν και ξανανοίγει με αίτηση ενός βουλευτή που δεν ανήκει στην Επιτροπή μας, αλλά φυσικά κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει να υπάρξει και πάλι αίτηση για άνοιγμα και πάλι μιας ε, αναφοράς. Αφού όμως είδα αυτή την αίτηση και είδα τις, ε, την αιτιολόγηση που έδωσε αυτός ο βουλευτής, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι μονάχα να επαναλάβω αυτό που είχαμε πει στο παρελθόν, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για να ανοίξει και πάλι αυτή η η αναφορά. Και αν λοιπόν συμφωνείτε θα ήθελα να ζητήσω να υπάρξει μια ψηφοφορία στην Επιτροπή μας όπου η ομάδα του ΕΛΚ θα ψηφίσει κατά του να ανοίξει και πάλι αυτή η αναφορά. Οι παρόντες συνάδελφοι θέλουν να τοποθετηθούν όσον αφορά το αίτημα του συναδέλφου Ιτουργάης. Allora, votiamo la, la richiesta... Ψηφίζουμε το αίτημα του συναδέλφου Ιτουργάη να μην ξαναανοίξει, να αφήσουμε κλειστή λοιπόν αυτή την αναφορά, την αναφορά 481 του 2009. Ποιο είναι υπέρ? Κατά αποχέ. Οπότε αποφασίζουμε να μην ξανανοίξει αυτή η αναφορά. Υπήρξε και άλλη ανακοίνωση που ήθελα να σας κάνω που συμφωνεί με αυτή και η κυρία Όκεν που δεν είναι παρούσα όσον αφορά τα αποτελέσματα της συνάντησης του Διαμασολοβητού του Ευρωπαίου, με τον Ευρωπαίο Διαμασολοβητή στην Κοπενχάγη. Εκεί συμμετείχε η αντιπροσωπεία της Επιτροπής, κυρία Όκεν. Θα ζητήσουμε αν θέλει να μας περιγράψει κάποια πράγματα στη συνέχεια των εργασιών της Επιτροπής μας. Πάω λοιπόν τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας ε, διάταξης. Έχουμε την 396 του 2009 που παρουσιάστηκε από τον κύριο Φατώνε, Ιταλό επίκο, με 152 υπογραφές και έχει σαν στόχο την εγκατάσταση μονάδας εξεργασίας λιμάτων στην περιοχή Κούμα Λίκολα στην Ιταλία. Ο αναφερόμενος δεν είναι παρόν. Οπότε, ως συνήθως, δίνουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Γιουζέπε Μαγκανάρο. Καλημέρα. Αυτή η εγκατάσταση υπεξεργασίας λιμάτων της ΚΟΥΜΑ είναι τώρα αντικείμενο δύο έρευνών που έχουν δρομολογηθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται η έρευνα όσον αφορά τη συμβατότητα αυτής της εγκατάστασης με την οδηγία όσον αφορά την εξεργασία των λιμάτων την 91-271 ε, παραβίαση του άρθρου 3 και του άρθρου 4 εικάζεται ότι έχουν συμβεί της οδηγίας. Το άρθρο 3 προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν επαρκή συστήμα αποχέτευσης για την συλλογή αυτών των ε, αποβλήτων και το άρθρο 4 προβλέπει ότι τα λύματα θα, που μπαίνουν στο σύστημα αποχέτευσης θα πρέπει να υπόκειται σε επαρκή κατεργασία. Οπότε χρειάζεται να υπάρχουν εξεργασίες λιμάτων που ε, πληρούν κάποιες προδιαγραφές ε, τεχνικές. Όσον αφορά αυτή την εγκατάσταση, τη ΚΟΥΜΑ, πάνω απ' όλα καλύπτεται από τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τις διοικητικές παραδιάσεις του, 2000, του 2034 έχει προτείνει ήδη προσφυγή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δηλαδή τελούμεν αναμονή της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που θα μας πει αν και για αυτή την εγκατάσταση της Κούμα από πλευράς των Ιταλικών αρχών έχει παραβιαστεί το άρθρο 3 της οδηγίας όσον αφορά την συλλογή αυτών των λιμάτων και την παροχή στην αποχέτευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε κάποιες πληροφορίες που δείχνουν ότι ίσως σε σχέση με αυτή την εγκατάσταση της Κούμα, ίσως να υπάρχει και παραβίαση του άρθρου 4, δηλαδή επεξεργασία των λιμάτων, των υγρών λιμάτων, όσον αφορά τη δεύτερη ενδεχόμενη παραβίαση οδηγίας, ακόμα διενεργείται μια προκρατική έρευνα που αφορά πάνω από 400 ε, περιοχές αστικές στην Ιταλία. Είναι πολύ περίπλοκη η τεχνική προσέγγιση, δεν έχει ολοκληρωθεί. Όταν οι υπηρεσίες θα έχουν ολοκληρώσει την αξιολόγηση, ε, θα αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν. Πιθανότατα θα ξεκινήσει μια διαδικασία κατά παράβαση που θα αφορά συγκεκριμένα την παραβίαση του άρθρου 4 και πιθανότατα αν η αξιολόγηση τεχνική επιβεβαιώσει ότι πράγματι η εγκατάσταση της Κούμα παραβίασε και το άρθρο 4, η εγκατάσταση της Κούμα θα καλύπτεται από αυτή τη νέα διαδικασία παράβασης. Εν τω μεταξύ, οι Ιταλικές ε, αρχές εστράφησαν προς τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ζήτησαν συγχρηματοδότηση για ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων και της παράβασης όσον αφορά την εγκατάσταση της Κούμα, οι Ιταλικές αρχές ζήτησαν συγχρηματοδότηση ενός προγράμματος ε, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αξιοποίησης ε, των διαφόρων υδάτων της περιοχής που είναι κάτι που ε, όσον αφορά και τα υπόγεια υδάτα που αφορά και την εγκατάσταση αυτή της Κούμα γίνεται αξιολόγηση πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το αίτημα των Ιταλικών αρχών δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αλλά υπάρχει και η δυνατότητα αυτή η τελευταία πρωτοβουλία να συμβάλλει τελικά ε, στην κάλυψη αυτής της παράβασης, στην, στην αυτή η παράβαση, να εξισορροπηθεί. Ζητά κάποιος να πάρει το λόγο, κάποιος συνάδελφος. Μποστινάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. As long as the commission... Όσο η Επιτροπή μας διαβεβαιώ, διαβεβαιεί ότι υπάρχουν προβλήματα και μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση. Εμείς θα πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά και πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή να μας κρατήσει ενήμερους σε σχέση με τις εξελίξεις και τα συμπεράσματά της και μπορούμε ενδεχομένω να οργανώσουμε εάν απαραίτητο και μία άλλη συνάντηση για τα θέματα αυτά. Είναι σαφές όμως ότι υπάρχουν προβλήματα, γι' αυτό εγώ πιστεύω θα πρέπει να παραμείνουμε ε, επάγρυπνη και να παρακολουθήσουμε την ενημέρωση της Κομισιόν. Το θέμα αυτό δεν είναι πια σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών, σε επίπεδο επιτροπής η οποία παρακολουθεί τη σύνολη διαδικασία και τις εξελίξεις. Και εγώ έχω την ίδια αντιμετώπιση, ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή δηλαδή η αναφορά. Η Κομισιόν μας είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια διαδικασία επί παραβιάση αλλά επίσης μας είπε η Κομισιόν ότι από την πλευρά των ε, Ιταλικών αρχών γίνονται προσπάθειες να υπάρξουν επενδύσεις και χρηματοδότηση για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Αυτό είναι καλύτερο λοιπόν γιατί δεν αρκεί να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι πολύ καλύτερο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και είναι θετικό ότι υπάρχει μια τέτοια κίνηση από την πλευρά των αρχών. Καταρχήν λοιπόν γίνεται η αναγνώριση του προβλήματος και δεύτερον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 Δίνω το λόγο στον ε, αρμόδιο της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εξ ονόματος Κομισιόν να σας πω ότι πράγματι απευθύνθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου μια όχληση προς την Ιταλία του 2011. Στις 13 Οκτωβρίου υπήρξε αιτιολογημένη γνώμη πήραμε τις ε, συμπληρωματικές πληροφορίες σε σχέση με ορισμένα σημεία της αναφοράς αυτής για θέματα τα οποία είχε αναφέρει ο αναφερόμενος στο παρελθόν αλλά δεν είχαν συμπεριληφθεί στην όχληση για λόγους που αναφέρονται και στην επιστολή της 30ης ε, Νοεμβρίου του 2010. Οι πρόσθετες αυτές πληροφορίες που ήρθαν σε γνώση μας πρόσφατα αφορούν αυτά τα σημεία βέβαια που είχαν αγερθεί προηγουμένω. Η Κομισιόν θα αναλύσει αυτά τα σημεία και θα πρέπει να υπάρξει πλήρης εξέταση αυτού του εγγράφου επειδή είναι 70 σελίδων και πέραν το έγγραφο αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει να περατωθεί μάλλον η μετάφρασή του και μετά να αρχίσει η ανάλυση για να δούμε κατά πόσον η Κομισιόν θα αναθεωρήσει τη στάση της και τα συμπεράσματα αυτά τα οποία είχε, στα οποία είχε καταλήξει, αν θα χρειαστεί να τα αναθεωρήσει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον αναφερόμενο για τις περαιτέρω πληροφορίες που μας έδωσε σε σχέση με την κατάσταση στην Ιταλία. Κάποιος θέλει να λάβει τώρα τους συναδέλφους. Αν κατάλαβα καλά, η Κομισιόν Ε, είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ένα διάλογο. Υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία που δόθηκαν από τον αναφερόμενο, τα ελέγχει η Κομισιόν και ζητά περαιτέρω στοιχεία από την Ιταλική κυβέρνηση και στο τέλος θα υπάρξει και πάλι μια εξέταση του κατά πόσο έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα από την Ιταλική πλευρά. Αυτή είναι η κατανόησή μου, δηλαδή στο τωρινό αυτό στάδιο εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε μια οριστική απάντηση κατά 100%. Γι' αυτό θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιό να μας κρατήσει ενήμερους μόλις έχει περαιτέρω στοιχεία και όταν υπάρξει μια τελική απόλυξη στο διάλογο μεταξύ των Ιταλικών αρχών και της ε, Κομισιόν. Δεν μπορούμε εμείς να εμποδίσουμε τη συνέχιση της συζήτησης. Ο κύριος Μποστινάρου. θέμα της αναφοράς αυτής. Θα ήθελα να σας διευκρινίσω ότι πρόκειται για απλώς την πρώτη καταχρονική σειρά από αυτές τις αναφορές την οποία τώρα διεκπεριώνουμε. Η προβληματική εδώ είναι πάρα πολύ τραγική από πλευρά ενό κράτου μέλου. Όμω δεν είναι εδώ μία μεμονωμένη περίπτωση. Διότι και στη δική μου χώρα, την Ρουμανία, ο αριθμό των ε, εργατικών ατυχημάτων έχει αυξηθεί ενισχυτικά. Και μετά τον αριθμό των θυμάτων των τροχαίων σε πολλά κράτη-μέλη είναι πόλεμο. Γιατί πάρα πολλοί ε, κόσμος πεθαίνει λόγω της έλλειψης ασφάλειας στην δουλειά. Οι εργοδότες δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στη δουλειά. Ούτε τιμωρούνται οι υπεύθυνοι όταν έχουμε τέτοια ατυχήματα. Δεν πρόκειται μόνο για τους εποχιακούς. Για αυτούς που έχουν τα σχετικές συμβάσεις εργασίας, ούτε μόνο για τους λαθρομετανάστες. Εδώ έχουμε να κάνουμε με εργαζομένους κανονικούς, οι οποίοι έτσι έχασαν τη ζωή του και πολλέ φορέ είναι συμβολικού χαρακτήρα η ευθύνη που αποδίδεται ει του εργοδότες. Επομένως θα πρέπει να ανακρούσουν τον κώδικα του κινδύνου. Και εγώ αλλά και η πολιτική ομάδα θέλουμε να απευθυνθούμε σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τη ζητήσουμε. Να μπορέσει να κάτσει και να κάνει μια πραγματική εξελίξη του τι κατάσταση επικρατεί στα κράτη-μέλη. Και κυρίω τώρα που περνάμε την περίοδο τη κρίση, διότι, διότι, διότι, στον βωμό του μαμονά κάνουν ό,τι να είναι. Οι τόσο έτσι να συμπιέσουν το κόστο. Δεν κάνουν τίποτα δηλαδή για την πρόληψη των αντιγνώτων οπότε και οι εργαζόμενοι έτσι ε, εξωθούνται να κάνουν ό,τι μπορούν. Όμω θα έπρεπε λοιπόν, να του εξωθήσουμε του εργοδότε να κάνουν ό,τι μπορούν για να έχουμε πρόληψη των ατυχημάτων. Επομένω, επομένως, προσοχή. Προσοχή διότι οι επίσημε στατιστικές πολλέ φορέ είναι αναλυθείς. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάτσει και να ανοίξει διάλογο με τα συνδικάτα. Να δει τα στοιχεία εκείνων και να δει κατά πόσο αντιστοιχούν τα στοιχεία των συνδικάτων με τα επίσημα στοιχεία. Και να δούμε επιτέλου τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο ώστε να μπορέσει να αντιδράσει δυναμικά. Να δείξει πυγμή. Και έτσι οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη να μην δουλεύουν σε καταστάσεις και συνήθω όπω οι Κινέζοι. Βεβαίω και να προστασία και κοινή. Όμω πολλέ φορέ ε, έχουμε το ίδιο άσχημε συνθήκε εργασία όπω και στην Κίνα. Επομένω θα μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και περιμένουμε να δούμε τι συνέχεια θα δώσει η, ε, σε επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παίρνουμε επίση περιμένουμε και κάποια ενημέρωση από πλευρά συνομοσπονδία ε, εργαζομένων <clears throat> και των πλευρά μελών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα θέλει ήδη να δώσει κάποιες απαντήσεις στα τεθέντα ερωτήματα. Peut-être juste, peut juste une chose, cette mise en demeure contre l'Italie, ça prouve que la Commission... Αυτή κατηγορία προς την Ιταλία επιβεβαιώνει το ότι η Επιτροπή είναι φιλικά των συνθηκών, όπως προβλέπετε. Δεν μπορούμε ακόμα να καταλήξουμε για το κατά πόσον είχαμε παραβιάσει τις συνθήκες, ούτε γι' αυτό έχουμε αυτήν την όχληση, την προειδοποίηση προς την ε, Ιταλία. Φυσικά και δεν στερείται μέσα στη όμως αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει το καθήκον της. Υπάρχει στρατηγική όσον αφορά την ασφάλεια στον χώρο εργασία και αυτό αποδίδει αποτελέσματα και έχουμε αναπτύξει και πρωτοβουλίε που βρίσκονται τώρα να εξελίξει. Σα ευχαριστώ. Και αυτοί και παρόμοιε αναφορέ χρονολογείται από το 2009. Πέρασε κάποιος χρόνος. Και εδώ μιλάμε για μη συμμόρφωση όσον αφορά την ομοθεσια Όχι μη επαρκή εφαρμογή που ίσως απαιτούσε έρευνα ενδελεχέστερη για αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Ελπίζω να προχωρήσουν οι εργασίες. Εν πάση περιπτώσει θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά για να δούμε ποιες εξελίξεις υπάρχουν μετά από την επιστολή με την όχληση και ποια θα είναι τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις όσες πληροφορίες που απεστάλησαν από τον αναφέροντα. Θέλει να απαντήσει ο αναφέρον. Δεν υπάρχει τίποτα που ήθελα να πω, παρατηρείται όμως ότι οι νεκροί ή τα τυχήματα που συνέβησαν στην Ιταλία υποεκτιμούνται πολύ, υποτιμούνται πολύ. Τα επίσημα στοιχεία είναι το είναι του Εθνικού Ινστιτούτου του αρμόδιου φορέα. Λαμβάνει υπόψη μόνο τους ασφαλισμένους, όχι τους μη νόμιμους εργαζομένους και υπάρχουν πολύ πολύ πολύ άλλοι ακόμα. Σε αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να προσθεθούν τουλάχιστον άλλοι 200 θάνατοι και όχι μόνο. Λάβετε υπόψη ότι κάθε μέρα πεθαίνουν δύο-τρία άτομα και σε κάποιες, κάποιες μέρες πεθαίνουν ε, πέντε, πάνω από πέντε άτομα και δεν είναι όλοι οι Ιταλοί που πεθαίνουν στα ατυχήματα. Ευχαριστώ. Ελπίζουμε πιο γρήγορη εξέλιξη όσον αφορά τις όλες διαδικασίες από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάμε στην αναφορά του επομένου σημείου, που είναι η 1153 του 2009, του κυρίου Τζίνο Τρεβιζανάτο. Είναι το σημείο στο οποίο πήγα λάθος πριν. Δίνω το λόγο στον αναφέροντα, που είναι παρόν. Ο κύριος λοιπόν Τρεβιζανάτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής των Αναφορών. Σας ευχαριστώ διότι μου δίνετε την ευκαιρία να σας αναπτύξω τα θέματα της αναφοράς μου κατόπιν του της ενημέρωσης που μας παρέσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω ότι όσα θα σας πω πρόκειται να οδηγήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διακόπτη ο μιλητής διότι σβήνει το μικρόφωνο του. Τώρα έρχεται, σας έρχεται. Α, μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν ότι εδώ μέσα για μια κατηγορία ζωμένη στην Ιταλία, οι οποίοι νομίζω έχουν τα ίδια ε, δικαιώματα όπω και άλλε κατηγορίε σε σχέση με τι ε, διατάξει που ισχύουν όσον αφορά τι ομαδικέ απολύσει. Και όπω θα προκύψει, χρειάζεται να εκδοθεί δεσμευτική απόφαση του σε ΟΚ, ούτω ώστε να κατησχίσει το κοινωτικό δίκαιο σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα πολιτών και εργαζομένων. Αυτό πηγάζει από το δικαίωμα στην προστασία κατά και σβήνει πάλι το μικρόφωνο μιλητή. Α, τώρα λειτουργεί, αλλά μόνο το έσβησε πριν. Και... Τα στελέχη είναι άνθρωποι ορχήστρα. Μιλάμε τώρα για κάποιους που στην IBM δεν συμμετέχουν στη δικασία στη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 1 της οδηγίας όσον αφορά κάποιες διαβουλεύσεις για να υπάρχουν κάποιο είδους ε, υπεράριθμοι εργαζόμενοι και αυτό οδηγεί σε κάποιες ομαδικές απολύσεις και οι λόγοι που επικαλούνται τέλο πάντων δεν περνάνε μέσα σε διαβούλευση και υπάρχει ατιώδη συνάφεια με αυτά που ε, επιχειρήματα έχουν να πούνε οι εργαζόμενοι. Οπότε έχουμε τώρα αυτή την οδηγία. Αυτή μεταφέρει στο δίκαιο του 1991. Πρόκειται για την πρώτη οδηγία σε σχέση με αυτό. Αλλά είχαν προηγηθεί και άλλε οδηγίε, η πρώτη εκ των οποίων ε, ανάγεται στο 75. Οπότε η δράση στο ιστορικό δίκαιο ξεκίνησε το 2010. Τότε το ακυρωτικό τη Ρώμη εξέδωσε μία απόφαση και είπε ότι η έφεσή μου είναι απαράδεκτη ε, κατά της απόφασης του δικαστηρίου του Μιλάνου διότι δεν ίσχυσε η αρχή της, ε, της έμεσης ισχύω της ε, οδηγίας. Και αυτά τα διευθυντικά στελέχη τελικά δεν ευεργετήθηκαν από τις ε, διατάξεις του σχετικού νόμου και νομίζω ότι τον Ιούλιο του 2007 μετά την απόφαση του ακυρωτικού ή του εφετείου εγώ προσέφερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι ξεκίνησα ε, αυτές τις δύο αναφορές και κατόπιν ξεκίνησε η διαδικασία παραβάση κατασταλής από προβάση της Κομισιόν. Οπότε, το θέμα εδώ δεν απαιτεί εφαρμοστικά μέτρα, αλλά το ερώτημα το οποίο υπέβαλα έχει ως εξή. Δεν θα έπρεπε η οδηγία για τις ομαδικές απολύσεις να παράσχει την ε, ίδια προστασία εις όλες τις κατηγορίες Ιταλών εργαζομένων δεδομένου ότι η διάταξη του πρώτου άρθρου αλλά και η ερμηνεία αυτού όπως προέκυψε εις δύο αποφάσεις του ΔΕΚ λένε ότι κατησχεί το κοινοτικό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο, το οποίο σε μερικέ περιπτώσει εξέρχεται από από την αφορμή αυτού του άρθρου. Επίση, το ακυρωτικό ή το εφετείο είπε για το παράδειγμα ότι από τότε που, που τέθησε ισχύ ο νόμος 2003 του 1991 αυτός κατησχύει όσον αφορά τις συλλογικέ απολύσεις. Πέρασαν 7 χρόνια και άλλα 4 τότε που εγώ άρχισα τον αγώνα μου. Όμως ακόμα ακόμα ε, δεν ισχύει η αρχή του κράτους δικαίου όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις αυτών των διευθυντικών σταλαγών και από το ανώτατο δικαστήριο δεν υπάρχει κάποια, ε, κάποιος κανόνας ούτε και από την ΙΟΚ. Θα έπρεπε όμως να έχει μεταφερθεί στο στρατό δίκαιο η σχετική οδηγία. Σαφώς προκύπτουν τα εξής. Πρώτον, δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν οι συλλογικές απολύσεις σε ατομικές. Επί τη βάση της νομολογίας αυτού του Ιταλικό και επίση. επίσης. Δεν είναι δυνατόν να προβαίνουν σε αυτές τις ε, ομαδικές απολύσεις μόνο κατά διευθυντικών στελεχών κάποιοι όπως η IBM. Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουν τα κεκτημένα δικαιώματα μια μερίδα μόνο των εργαζομένων όταν κάποιες εταιρείε έχουν πάνω από 15 εργαζομένους προσλαμβάνουν τα δύο τρίτα των εργαζομένων στην Ιταλία και έτσι αποκλείουν τις προστασίες του νόμου 223 προς τους υπεράριθμους όλων των κατηγοριών και οπότε θα έπρεπε να, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το κατόφλι των πέντε εργαζομένων σε συγκεκριμένες μέρες που ο νόμος και αυτό το κάνουν χωρίς να υπολογίζουν τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών στο, σε αυτόν τον αριθμό για τη διάταξη αυτή της προθεσμίας. Δεν είναι εφαρμοσμό την, ε, την οδηγία για τα διευθυντικά στελέχη. Έχουμε την απόφαση 78 του 80. Θα έπρεπε αυτό να το σεβαστεί το Ιταλικό ακυρωτικό. Όμως, επικαλέστηκε κάποιες ατομικές απολύσεις. Το εταιρικό κυρωτικό λόγω σφαλμάτων, λόγω ανεπαρκής των εργαζομένων. Επομένως. Επικρατεί μια έλλειψη ασφάλειας δικαίας των τελικά των αυτών. Αυτό προβλέπει τα δικά μου συμφέροντα. Αυτός ο δικός αγώνας μου επέφερε μεγάλη ζημία, αλλά έτσι, παραβιάζει το άρθρο 30 η Ιταλία στον αφορά την προστασία κατά των δικαιολογικών απολύσεων, το άρθρο 27 στον αφορά τα δικαιώματα των εργαζόμενων στη διαβουλή, το άρθρο 41 το οποίο είναι το δικαίωμα στην χρηστή και δίκαιη διοίκηση και επίση το 47 όσον αφορά την, ε, το δικαίωμα ή στα ένδικα δικαιώματα και, θα, και στην προσφυγή ή στο χάρτη των θεμελιών δικαιωμάτων, γιατί εκεί έχουμε το άρθρο 51 το οποίο μπορεί να το επικαλεστεί και θεσμικό όργανο, μπορεί να σου πει και κράτο μέλο Κάθε Οπότε, εν κατακλείδη, θα πρέπει να έχουμε μια δεσμευτική απόφαση τη ΙΟΚ σε σχέση με την ε, συζήτηση αναφοράς. Ε, και θα πρέπει να δοθεί σωστή απάντηση και να δοθεί απάντηση αυτό που ερώτησα. Ε, κατηγορούν, ε, ε, καλύπτονται ή όχι από το πεδίο εφαρμογή αυτή τη οδηγία του Συμβουλίου τα διευθυντικά στελέχη όσον αφορά τι συλλογικέ απολύσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κ. Δημήτρη Δημητρίου. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω πρώτα απ' όλα ότι επειδή ότι μετά από την ανακοίνωση της Κομισιόν τον Ιούνιο του 2011 η Κομισιόν έστειλε και στην, στην Ιταλία μια συμπληρωματική επιστολή προειδοποίησης όχλησης και η Κομισιόν ήθελε με την επιστολή αυτή να συγκεκριμενοποιηθούν αυτές οι καταγγελίες που περιλαμβανόντουσαν ήδη στην πρώτη επιστολή όχλησης. Οι Ιταλικές αρχές είχαν απαντήσει σε προηγούμενες επιστολές και χρειαζόμασταν να εξετάσουμε τα στοιχεία αυτά, γι' αυτό ζητήσαμε περαιτέρω διευκρινήσει προς το τέλος Σεπτεμβρίου, <clears throat> στις 30 Σεπτεμβρίου, πιο συγκεκριμένα του 2011, του ενεστώτους έτους. Στη συνέχεια επίσης αναφερθήκαμε και απευθύναμε και προς τον αναφερόμενο μία επιστολή στα τέλη Οκτωβρίου του 2011, όπου πληροφορούσαμε λεπτομεριακά τον αναφερόμενο για τις λεπτομεριακά για τις εξελίξεις και για το περιεχόμενο των προσφάτων επιστολών της Κομισιόν προς τις Ιταλικές Αρχές. Για να απαντήσω λοιπόν στον αναφερόμενο, πρώτα απ' όλα θέλω να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία του με τις υπηρεσίες της Κομισιόν και τις πληροφορίες που έφερε εις γνώση μας. Και δεύτερον, να απαντήσω ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συμπληρωματική επιστολή όχλησης υπέδειξε στις Ιταλικές Αρχές <clears throat> ότι οι dirigenti, η κατηγορία λοιπόν αυτή των στελεχών, εξαιρούνται από την εμβέλεια εφαρμογής του Ιταλικού νόμου, ο οποίος έχει σαν ε, στόχο να μεταγράψει την αρμόδια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κομισιόν υπογραμμίζει το γεγονός ότι κατά την άποψή της η Ιταλία παραβιάζει τις ε, απαιτήσεις της οδηγίας. Έχουν τώρα λοιπόν δύο μήνες οι Ιταλικές αρχές μετά από την αποστολή αυτής της ε, επιστολής να απαντήσουν. Έχουν ακόμα ένα μήνα για να απαντήσουν. Και φυσικά θα δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες στην Επιτροπή σας και στον αναφερόμενο για τις εξελίξεις που θα προέλθουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο, ο κ. Μποστινάρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φαίνεται ότι σήμερα οι Ιταλοί, οι Ιταλοί αναφερόμενοι επεκτείνονται σε νέους χώρους αναφορών. Αυτό δείχνει ότι αυξάνουν τα προβλήματα στην Ευρώπη μας και αυξάνει και η απόγνωση του πληθυσμού. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρξει όχι μονάχα στα χαρτιά, αλλά και στην πραγματικότητα. Γιατί σας τα λέω αυτά, γιατί όλα αυτά δεν αφορούν μονάχα την Ιταλία. Δεν αφορούν τα συλλογικά δικαιωμάτια των εργαζομένων στην Ιταλία. Πρόκειται για μια διαδικασία επιμόλυνσης και άλλων κρατών μελών εν εξελίξει. Όπως ξέρετε, κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν αλλάξει οι εργασιακοί κώδικες και σε άλλες χώρες, στην Ρουμανία και στην Ουγγαρία συγκεκριμένα. Και ίσως ξέρετε ότι μέσα στο νέο εργασιακό αυτοκώδικα που ενεκρίθη το 2011, τουλάχιστον στην περίπτωση της Ρουμανίας, η οποία αντικατοπτρίζει τα τεκτενόμενα στην Ιταλία. Δεν υπάρχει δυνατότητα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δεν υπάρχουν ε, εθνικές συλλογικές συμβάσεις και ο εργοδότης δεν έχει καν την ανάγκη για να εξηγήσει γιατί απολύει κάποιους. Τίποτα, μηδέν. Ξαναγυρίζουμε στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτή είναι μια δραματική εξέλιξη και πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αφορά αυτό μοναχά τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες συνήθως έχουν μια τέτοιου είδους συμπεριφορά που στρέφεται κατά των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ευρώπη. Ακόμα και εγχώριες μικρές εταιρείες ακολουθούν την εργασιακή πολιτική των μεγάλων εταιριών, των μεγάλων πολυεθνικών. Και το 2008 η Νόκια αποφάσισε να κλείσει το εργοστάσιο της στη Μπόχουμ. Ο συνάδελφος θα μπορούσε να το επιθυμήσει. Αυτό έγινε με σημαντικές αποζημιώσεις για τους Γερμανούς εργαζόμενους που απελήθησαν συλλογικά. Όταν όμως υπήρξε μια αντίστοιχη κατάσταση στη Ρουμανία, η ίδια εταιρεία η Νόκια έκλεισε το εργοστάσιο στην Κλούσνα με αποζημίωση της τάξης των 6 ή 8 μισθών, μιλάμε για 200-250 ευρώ το μήνα, επειδή ο νέος κώδικας εργασίας που έχει εγκριθεί στη Ρουμανία, που αντιβαίνει με την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη θέση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στην Ευρώπη, επιτρέπει στη Ρουμανία επιτρέπεται παρόλα αυτά στη Ρουμανία να εφαρμοστεί ένας τέτοιος κώδικας. Και αναφέρομαι και στον Ιταλό αναφερόμενο, θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι τώρα υποσκάπτουμε την κοινωνική βάση της Ευρωπαϊκή μοντέλο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξακολουθούμε να παριστάνουμε ότι έχουμε ένα κοινωνικό μοντέλο, το οποίο όμως ουσιαστικά είναι υποεξαφάνιση. Στη μέση της κρίσης αυτής της χρηματοπιστωτικής είναι καθήκον της Κομισιόν να αναλάβει δράση εναντίον τέτοιων πρακτικών, να τη σταματήσει και να επανορθώσει την κατάσταση εάν θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες να εξακολουθούν να πιστεύουν ότι υπάρχει κοινωνικό υπόδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ δεν μιλώ ως κάποιος ο οποίος είναι από την αριστερή πολιτική πτέρυγα, ως, αλλά ως κάποιος που ενδιαφέρεται για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αντιμετωπίζουμε έτσι τους εργαζομένους, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να υποσκάψουμε την ε, έννοια της Ευρώπης και να καταρακώσουμε την σταθερότητα και την αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ λοιπόν, λέει στον αναφερόμενο κύριο Μποστινάρου. Σας ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Ο κύριος Γιάρεκ έχει το λόγο. Äh, Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες ε, γενικές διαπιστώσεις. Αυτά που βλέπουμε είναι και αυτά ένα κομμάτι μιας Ευρώπης που εξακολουθεί να είναι ακόμα ζωντανή ενώ τις αναφορές οι οποίες ε, υποβάλλονται εδώ. Η, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο κάνουν την νομοθεσία. Οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν εμπιστοσύνη ότι αυτή η νομοθεσία θα εφαρμοστεί και έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται και να καταγγέλνουν όταν δεν υπάρχει η σωστή μεταγραφή αυτής της νομοθεσίας στην, ε, στη χώρα τους. Αυτό είναι λοιπόν ένα από τα κεντρικά σημεία της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μπορεί να μην έχουμε σε ορισμένε περιπτώσει νομοθεσία, αλλά όταν υπάρχει νομοθεσία υπάρχει κάθε δικαίωμα του πολίτη να ζητήσει να εφαρμόσουν σωστά αυτά τα, αυτές οι νομοθεσίες. Ίσως θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με τις αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπές. Να, για να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να παρακολουθούμε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, κάνουμε, εκδίδουμε κάποιους νόμους, αλλά δεν έχουμε κανένα τρόπο να ελέγξουμε πώς γίνεται η μεταγραφή και η εφαρμογή των νόμων στα κράτη-μέλη. Έχουμε σε περίπτωση, ε, παραδείγματος χάρη, διατάξεων για την γεωργία, χρονικά διαστήματα μέχρι και 12 χρόνια για την πλήρη εφαρμογή αυτό το διατάξεων και παρόλα αυτά διαμαρτύρονται ορισμένα κράτη-μέλη ότι 12 χρόνια είναι πολύ γρήγορα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα καλύτερο τρόπο για να έχουμε μια ταχύτερη εφαρμογή όλων αυτών των ε, νομοθετημάτων, να μην έχουν τα κράτη-μέλη ένα απεριόριστο ουσιαστικά χρόνο για την εφαρμογή του στην πραγματικότητα και φυσικά μπορούν τα κράτη-μέλη πάντα να μας λένε αν έχουν κάποιο συγκεκριμένο χρόνο και όχι να περιμένουμε τους αναφερόμενους. Όλα αυτά σας τα λέω λιγάκι στο, σε αφηρημένο επίπεδο, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, δεν αρκεί λοιπόν η Κομισιόν απλώς να δίνει την εμπιστοσύνη της στα κρατημέλη. Τα κρατημέλη θα εφαρμόσουν σωστά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ζούμε σε ένα αγγελικό κόσμο. Τα κρατημέλη πολλές φορές ακολουθούν τη δική τους οδό και επομένως θα πρέπει να έχουμε και μια συζήτηση ενδεχομένως με την Νομική Επιτροπή για το πώς θα μπορέσουμε να βρούμε ένα καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων μέχρι να φτάσουμε σε το σημείο είναι απαραίτητη η λειτουργία της Επιτροπής Αναφορών και θέλω να ευχαριστήσω και τους αναφερόμενους οι οποίοι έρχονται ενώπιόν μας για να μας δείξουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Για τη συγκεκριμένη αναφορά βέβαια μας λείπουν ακόμα πληροφορίες, πρέπει να την κρατήσουμε ανοιχτή. <clears throat> Σας ζητώ όμως, ε, αναφέρομαι στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, να μας πληροφορήσετε το ταχύτερο δυνατό για τις εξελίξεις, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα, να δούμε αν υπάρχει πράγματι και μια διαδικασία επί παραβάση, την οποία θα ξεκινήσει η Κομισιόν στην περίπτωση αυτή. Θα ήταν λοιπόν απαραίτητο να υπάρξει και μια επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας και η Κομισιόν να υπενθυμίσει στα κράτη-μέλη ότι οι οδηγίες και οι κανονισμοί θα πρέπει να τηρούνται. Όλοι αυτοί οι κανονισμοί λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο προέρχεται εκ του ουρανού είναι αποφάσεις που έχουν ληφθεί με τη συνεργασία της Κομισιόν, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Τα κράτη-μέλη όμως δεν μπορούν να, δει, να παριστάνουν ότι δεν έχουν ιδέα όλα αυτά, γιατί έχουν αντιμετωπίσει αυτό το θέμα σε επίπεδο Συμβουλίου. Δεν μπορεί να μας λέει κάποιος ότι το αποφάσισαν οι Βρυξέλλες όταν ο ίδιος έχει συμμετάσχει στη διαμόρφωση των θέσεων των Βρυξελών. Με τέτοια παιχνίδια δεν μπορεί να λειτουργήσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν ανοιχτή αυτή την αναφορά και θέλω να ευχαριστήσω τον ε, αναφερόμενο για το γεγονός ότι δείχνει πόσο ζωντανή είναι ακόμα η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Δεν θέλουν άλλοι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο, νομίζω. Ο αναφέρον ε, θέλει να απαντήσει, να πει κάτι θα ήθελα να πω κάτι εν είδη ερωτήματος προς τον εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να μιλήσω ιταλικά, αγγλικά. Τι να μιλήσω. Θα με βοηθήσω να μιλήσω αγγλικά, διότι περισσότεροι παριστάμενοι ε, γνωρίζουν πιο καλά τη γλώσσα αυτή, τα αγγλικά. Ε, θα ήθελα να απευθυνθώ εις τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με αυτή την επιστολή προς τις τελικές αρχές. Μία από τις πιο πρόσφατες ή στις 30 ή 14 Σεπτεμβρίου. Και με αυτή τη δίμηνη προθεσμία μου τώρα όμως πέρασαν σχεδόν τρεις μήνες. Δεν πάμε μου λέτε εμένα ότι στείλατε τον Οκτώβριο και ακόμα δεν έχει φτάσει απάντηση από την Ιταλία. 21 Νοεμβρίου σήμερα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για το τι ισχύει σήμερα. Eh, είναι ένα ερώτημα που είναι απαντά από μόνο του νομίζω. Ακούγοντας τις προτάσεις των διαφόρων ε, συναδέλφων που μίλησαν, θα πρέπει, πιστεύω, να κρατήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά αυτή. Ευχαριστούμε τον αναφέροντο και που έθεσε δύο σημαντικές υποθέσεις και ίσως προκύψει και ο δέον προβληματισμός και στη συζήτηση των συντονιστών της Επιτροπής. Μπορεί να εντοπίσουμε μηχανισμούς και διαδικασίες που θα επιτρέψουν Επιτροπή Αναφορών να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα σε παρόμοιες περιπτώσεις. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω, όπως έλεγε και ο Πίτερ Γιάρ, να, δίνουμε χαρακ... να δώσουμε χαρακτήρα κατεπήγοντος και σημασίας και σε αυτή και στην προηγουμένη αναφορά, ε, να το προωθήσουμε στην Επιτροπή Εργασίας, να ζητήσουμε γνωμοδότηση, να αξιολογήσει το θέμα επί της ουσίας και να ξεκινήσει κάποια διαδικασία, κάποια διεργασία επί των τεθέντων ερωτημάτων. Όπω λέει και Μποστινάρο, αυτά τα θέματα δεν αφορούν μόνο την Ιταλία, αλλά πολλέ άλλε χώρε τη Ένωση. Άρα θα ήταν χρήσιμο να προσέξουμε αυτά τα σημεία. Ευχαριστώ και πάλι τον αναφέροντα. Πάμε στην επόμενη αναφορά, την 1557 του 2009. Υπευλήθη από την κυρία Ζαμπέλα Μεζάροσνη Γεωργάρη, Ουγγρικής Ιθαγένειας εξ ονόματος της Ένωσης για την Προστασία των Συμφερόντων των Επιχειρήσεων σχετικά με διακρίσεις σε βάρος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ουγγαρία και τη συμμόρφωση προς πρότυπα ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι αναφέρουσα παρούσα και τη δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μου δίνετε σήμερα ευκαιρία να σας ομιλήσω και σε αυτό το λίγο χρόνο που έχω θα ήθελα να σας φωτίσω ορισμένα θέματα τα οποία δεν διευκρινίζονται στο αρχικό έγγραφο. Δεν είναι ότι έχουμε αυτό το ποσοστό των απασχολημένων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 95% λέει το 2009, τα δύο τρίτα των εργαζομένων ήταν σε αυτόν τον κλάδο. Όμω, δεν του πρόσεξε και πολύ η κυβέρνηση. Όλε οι παραγωγικέ επιχειρήσει βρίσκονται σε παραγωγική κατάσταση. Ένα δισεκατομμύριο φιωρίνια βρίσκονται οι περίμερε οφειλέ. Δεν ο μιλητή, δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα τεχνικό, διακόπτη. Και έχουμε τώρα κάποιες ε, αθέμητες πρακτικές που έχουν οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες. Οπότε δεν καταβάλλονται κάποιες οφειλές ε, Οπότε θα πρέπει να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, όμως δεν βοηθούν οι αρχές οι οποίες δεν έχουν καμία ευελιξία και πολλές φορές έτσι τι συμφέρουν ακόμη περισσότερο διότι έχουμε μεγάλη γραφειοκρατία και βαριά φορολογία. Στην Αυστρία είναι τελείως άλλη υπόθεση σχέση επιχειρήσεων και αρχών. Οπότε δεν καταλαβαίνουν και οι αυστριακές επιχειρήσεις το πόσο άκαμπτο είναι το ουγγρικό σύστημα. Ακριβώ επειδή είναι έτσι δύσκολη κατάσταση, οι προοπτικέ είναι πάρα πολύ ζωφερέ. Έχουμε ιδιωτικό επίπεδο το οποίο πέφτει, έχουμε κοινωνική κρίση, έχουμε χρηματοοικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επίσης. Οπότε δεν υπάρχουν και πολλές ελπίδες ότι το κράτος θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Και οπότε το βάρος τώρα πέφτει στις ε, ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς ε, εντες εργασίας για να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Ε, δεν μπορεί το κράτος να διαφορεί για αυτές τις αθέμητες πρακτικές. Η χρηματοπιστωτική κρίση δεν γνωρίζει σύνορα. Οπότε έχουμε τέτοιες αρνητικές συνέπειες που υπονομεύουν και τις σχέσεις Ουγγαρίας με τους ε, μπουργούς τους εταίρους στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και πολλές επιχειρήσεις στη χώρα μας αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Αυστρία, στη Γερμανία, ή σε άλλες πιο αναπτυγμένες οικονομίες. Μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό 5 5-10 εργαζομένους. Υπάρχει όμως αρκετή εμπειρία, συστάσεις καλές και γι' αυτό και είναι επικερδής τα στριωτά τους, ακόμα και εκτός έδρας, στις ξένες αγορές. Όμως έχουμε αυτά τα φαινόμενα των αθεμήτων παγιών κυρίως από κάποιους ενδιάμεσους, αυτοί που μεσολαβούν μεταξύ των πελατών και αυτών των επιχειρήσεων. Δεν αποδίνουν αυτά που έπρεπε στην επιχείρηση. Όλα αυτά είναι άσχημα γιατί κλονίζει την εμπιστοσύνη των ε, επιχειρήσεων και έτσι υπονομεύει δραστηριότητά τους παρά το ότι βρίσκονται στα όρια της ε, χρεοκοπίας. Ούτε αυτό βοηθάει το μέλλον των νέων εργαζομένων, το οποίο είναι επίσης ζωφερό. Όμως, αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να τονωθεί η παραγωγικότητα. Έχουμε τώρα το 15 του Χάρτη των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, το οποίο ορίζει ότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται ίσων, ισοδυνάμων συνθηκών εργασίας. Από την μεριά έχουμε τι πολυεθνικέ. Εκείνε που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ουγγαρία. Και εκείνε. Αυτό το οποίο κάνουν είναι να ακολουθούν αυτέ τι αθέμητε πρακτικέ. Και παρακάμπτουν τι διατάξει και την νομοθεσία. Είναι παράδειγμα αυτή η κατάσταση. Είναι αφόρητη. Έχουμε τώρα το άρθρο 47 του Χαρτιδίου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τι ορίζει. Ότι όλοι οι Ευρωπαίοι δικαιούνται δικαστικής προστασίας και δικαίας δίκης. Πολλές φορές όμως δεν ισχύει αυτό το δικαίωμα στη χώρα μας. Δεν απονέμει τη δικαιοσύνη όπως θα έπρεπε. Οπότε και γι' αυτό έχουμε οικονομικές αρνητικές συνέπειες ηθικές συνέπειες και αφορά τους, αν, ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Είναι μακρές εφηγουρατικές διαδικασίες και αμφιβολά τα αποτελέσματα. Εμείς με ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε ότι οι ουγγρικές επιχειρήσεις έφτασαν τις συνέπειες της ανικανότητας της κυβέρνησης και της ανυπαρξίας υγιών συνδικών του επιχειρήν. Θα πρέπει να σταματήσει αυτού του είδους η, η ζημία βάρος τους. Αμελητή θα πρέπει να εφαρμοστούν τα όσα προβλέπονται από την νομοθεσία, τα δικαιώματά τους. Megtenni egy magyarral sem, különben az uniót létesítő alapelvek sérülnek. Tudjuk, hogy a magyar kormány súlyos örökséget kapott elődeitől, és a válság újabb Θα, έπρεπε και οι επιχειρήσει τη χώρα μα να απολαύουν των μάτων όπω και στην Πολωνία ή στην Γερμανία. Εντάξει, έχουμε τα μαρτύρια του παρελθόντο. Έχουμε επίση και την δυσμενή οικονομική σημερινή συγκυρία. Θα πρέπει να συγκρατήσει το χρέο η κυβέρνηση, να δώσει ανάπτυξη στην οικονομία. και να υπάρξει ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για τις ΜΜΕ. Και έτσι να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Εμείς περιμένουμε η Επιτροπή των Αναφόρων εδώ να σταθεί στο πλάι των δικαιωμάτων των ΜΜΕ και να έχουμε τέτοια δικαιώματα όπως χρειάζεται στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον Didier Μπουλού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κυρία Αναφέρουσα όσον αφορά το πρόβλημα που θέσατε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τις διάφορες καταγγελίες όσον αφορά το κοινοτικό δίκαιο. Το σημείο που υπογραμμίσατε είναι η σημασία που έχουν οι, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ουγγαρία, διαπιστώσαμε και το αναφέρουμε στο πρώτο μέρο τη απαντήσεις μα στο θέμα, αναφερθήκατε σε πέντε συγκεκριμένα σημεία όσον αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Το πρώτο σημείο μα επιστρέφει την προσοχή είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τι τράπεζε. Διαπιστώνεται ότι μονομερώ ε, τερματίζονται συμβάσει από τι τράπεζε. Σύμφωνα με το Δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, τα δάνεια που δίνονται στι επιχειρήσει δεν ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαραίτητα. Άρα τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόσει το δικό τους δίκαιο όσον αφορά ε, τα, τους όρους σύναψης δανείων με τις επιχειρήσεις σας και άλλο ε, θέμα. Το θέμα εκείνο που δεν πληρώνονται. Υπάρχει νομικό πλαίσιο μέσω της οδηγίας του 2011 του Φεβρουαρίου του 2016 όσον αφορά τι πληρωμέ και εκτέλεση πληρωμών για του προμηθευτέ. Υπάρχει αναρμόνιση τη περίοδου πληρωμών από πλευρά των δημοσίων αρχών προ επιχειρήσει, η συμβατική ελευθερία και όσον αφορά τι εμπορικέ συναλλαγέ το ότι επιχειρήσεις αυτομάτως έχουν την άδεια να ζητήσουν ε, τόκους για καθυστερήσεις πληρωμών και τα νόμιμα επιτόκια καθυστερήσεις πληρωμών ε, που δημιουργήθηκαν από τη νέα οδηγία για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος των ε, μη πληρωμών. Αν έχετε ανάγκη εξηγήσει συμπροματικές θα σας δώσουμε μετά όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο. Τρίτο σημείο που εφήγει αφορά ε, τους ε, των επιχειρήσεων. Υπάρχει διάκριση δηλαδή, στην εφαρμογή των, ε, της Ουγγρικής νομοθεσίας. Η οδηγία, η λογιστική απαιτεί δημόσιο, να έχουν αιτήσια λογιστικά οι διάφορες εταιρείε. Αυτό είναι αρμοδιότητα όμως των Ουγγρικών αρχών για τους κανόνες εφαρμόζονται. Άλλο σημείο αφορούσε τις δημόσιες προμήθειες και τα ερωτήματά σας όσον αφορά τις ε, προμήθειες αυτές. Θα θέλαμε καταρχάς να υπογραμμίσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, παίρνουν, ε, είναι ανάδοχοι των περισσότερων δημοσίων συμβάσεων, δίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναφέρεστε στι δημόσιε αυτέ αγορέ, δημόσιε προμήθειε, σαν μικρομεσαίε επιχειρήσει έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν στι ε, διαδικασίε αυτέ, στου διαγωνισμού αυτού. Καταρχά, να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα έγγραφο που δίνει κατευθυντήριε γραμμέ όσον αφορά το θέμα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και η οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ενώση όσον αφορά τι δημόσιε προμήθειε εμπεριέχει υποχρεωτικά κριτήρια αποκλεισμού. Παραδείγματο χάρη όταν υπάρχει περίπτωση διαφθορά και απάτη. Και άλλα κριτήρια που είναι σημαντικά για τον αποκλεισμό, όπω ε, διάφορα επαγγελματικά προβλήματα, έλλειψη κάποιων, μη πλήρωση κάποιων κριτηρίων και αυτά αντικαταπτρίζονται, το διαπιστώσαμε στον ελληνικό ε, νόμο, την αγγλική νομοθεσία όσον αφορά τι κρατικέ προμήθειε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δικασία παράβαση όταν ένα κάτω μέλο παραβιάζει κανόνε σχετικά με τι δημόσιε προμήθειε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τι δημόσιε προμήθειε ε, δεν βρήκε στοιχεία που να επιτρέπουν το να ξεκινήσει τη δικασία παράβαση. Όσον αφορά το κοινοτικό δίκαιο, αναφέρεστε μετά στη φορολόγηση. Και επικρίνεται η Ουγγρική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία οι αρχές μπορούν να ζητήσουν το ΦΠΑ όσον αφορά τι παραχόμενε υπηρεσίες όταν ε, δεν υπάρχει ε, συμβαλόμενο μέρο όσον αφορά παροχές. Σύμφωνα με τις οδηγίες για το κοινό σύστημα ΦΠΑ μπορεί να ζητηθεί πληρωμή φόρου τη στιγμή παράδοσης των αγαθών όταν η παροχή γίνεται ακόμα και αν η πληρωμή έχει αναβληθεί να πω εν κατακλείδη, εν συμπεράσματι, ότι είναι ενδιαφέρουσα η περίπτωσή σας, αλλά όπως είπατε η ίδια, δεν, δεν δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή της Ουγγρικής κυβερνήσεων ε, στο... και ότι είναι θύματα οι επιχειρήσει όσον αφορά την ανικανότητα του Ουγγρικού συστήματος. Δεν υπάρχει παραβίαση όμως του κοινοτικού δικαίου κατά την απόψή μας και για το θέμα αυτό αφορά αποκλειστικά, το εθνικό δίκαιο της Ουγγαρίας και αυτό έχω να πω αν ήδη απαντήσω στην αναφέρουσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Σταβάνα Μετ, στον συνάδελφο. Αν θέλετε να μιλήσετε για θέματα που άπτονται της ειδικότητάς σας, της αμμοδιότητάς σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να προσθέσω κάποια στοιχεία για την πολιτική σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ευθύνη της ε, Κομισιόν στα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να παρακολουθήσει και την πολιτική που ακολουθείται έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στα κράτη-μέλη. Είναι βέβαια εθνική αρμοδιότητα, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην Ουγγαρία και προσπαθούμε να επηρεάσουμε με θετικό τρόπο τις πολιτικές εναντί των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταρχήν με την νομοθεσία για τις μικρές επιχειρήσεις. Είμαστε επίσης σε, αρχές, σε συζητήσεις με τις εθνικές αρχές συγγνώμη, για την πολιτική ε, σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια της Ατζέντας 2020 και υπάρχει και ένα δίκτυο σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο κ. στην Ουγγαρία, είναι αυτός ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος για τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το δίκτυο αυτό των εκπροσώπων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συναντιέται τακτικά εδώ στις Βρυξέλλες για να συζητήσει τα θέματα της αρμοδιότητάς του, να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα προβλήματα και να υπάρξει και μεταλαμπάδευση εμπειριών και από ό,τι ξέρουμε και η τρέχουσα ουγγρική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει κάποια προγράμματα μέσω των οποίων θα αντιμετωπιστεί το διοικητικό άχθος και θα μειωθεί. Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά είναι ακόμα σε φάση εφαρμογής, επομένως οι επιχειρήσεις δεν μπορούν ακόμα να πάρουν τα θετικά στοιχεία αυτής της διαδικασίας, αλλά είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι οι κυβερνήσεις θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα. Δεν έχουμε άμεση δυνατότητα άσκησης πίεσης αλλά ξέρετε ότι εμέσως προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις ουγγρικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να κάνουμε την πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιο θετική σε όλη την Ευρώπη. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Η συνάδελφος άσκησε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να προβώ σε κάποια σύντομα σχόλια. Ναι, κυρία Χάνκης. Αυτή η αναφορά ανα... μιλάει για διάφορα προβλήματα που οδηγούν σε σοβαρές ανθρώπινες τραγωδίες. Αναφέρεται σε απλήρωτους λογαριασμούς και τη μη επιστροφή φόρου τη με αξίας. Δεν είναι ουγγρικό πρόβλημα αποκλειστικά. Αρκετά κρατημέλη έχουν μπροστά τους αυτά τα προβλήματα. Όσο περισσότερες χώρες πλήττονται από την κρίση κατά την άποψή μου, τόσο περισσότερο υποφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους. Διότι οι πολυεθνικές έχουν κεφάλαια να τις βοηθήσουν να βγουν από την κρίση, ενώ μικρομεσαίες επιχειρήσεις πέφτουν θύματα της κρίσης. Γι' αυτό είναι σημαντικό να το υπογραμμίσουμε το πρόβλημα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. να προσθέσω κάτι που ελπίζω να το δέχεται η αναφέρουσα. Θέλω να πω ότι δεν θεωρώ δίκαιο να αναφερόμαστε σε όλες τις κυβερνήσεις, ίσως για εκείνους που δεν γνωρίζουν την Ουγγαρία, θα έπρεπε να δείξουν ποιο είναι το πλαίσιο στη χώρα. Μετά από δύο τετραετίες σοσιαλιστικής κυβέρνησης, όπου υπήρξε αυτό το πρόβλημα, είδαμε ότι οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις ήταν κοινικές όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεν ασχολήθηκαν με τη θεμητή αυτή ανάγκη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από όταν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ουγγαρία, μόνο μια φορά μόνο μια φορά λέγω ήταν θύμα διαδικασίας παράβασης. Της απευθύνθηκε προειδοποίηση. Η παρούσα κυβέρνηση ανήκει στην οικογένεια του ΕΛΚ. Κληρονόμησε 100 δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια εξωτερικό χρέος. Αυτό ήταν αποτέλεσμα διαφόρων δημοσιονομικών προβλημάτων. Η παρούσα κυβέρνηση της χώρας έχει δηλώσει ότι είχε σαν πρωταρχικό στόχο την επίλυση των λόγω προβλήματος. Έγιναν διάφορα βήματα μέσω διαφόρων οικονομικών σχεδίων και προγραμμάτων. Η παρούσα κυβέρνηση κληρονόμησε επίσης μια συγκεκριμένη κατάσταση. Μια κατάσταση που πλησίαζε τη χρεοκοπία. Χρειάζεται συνεπώς χρόνος για να διορθωθεί η κατάσταση. Έχω και ένα υποκειμενικό σχόλιο. Δεν κατάγομαι από... Δεν προέρχομαι από κάποιο οικονομικό χώρο ε, και δεν έχω μεγάλες οικονομικές γνώσεις. Παρ' όλα αυτά θα εκφράσω μια άποψη. Διαβάζοντας την αναφορά, και έχοντα ερευνήσει το όλο ιστορικό της υπόθεσης και έχοντα ακούσει την αναφέρουσα και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ξέρω πώς να το πω αγγλικά, δεν ξέρω που στέκομαι όμω αυτό είναι το ζουμί. Δεν ξέρω που βρίσκομαι σαν αφορά την υπόθεση. Διότι αισθάνομαι ότι μιλάμε για πολλά ζητήματα που δεν νομίζω ότι αναφέρονται καν στην υποβληθής αναφορά. Διερωτώ με συνεπώς κατά πόσο μία λύση, αυτό το αποφασίζετε εσείς, προσπαθώ να βοηθήσω, κατά πόσο μία λύση, έλεγα, θα ήταν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και ενδεχομένως να ετοιμαστεί ένας κατάλογος που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους νόμους και τα νομικά μέσα που, όταν, που δείχνουν ότι δεν έχει συμμορφωθεί η Ουγγαρία με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι νομίζω ότι υπάρχει ουσιαστικό ζήτημα. και συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και μετά έχουμε άλλα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Νομίζω ότι περιέχονται κάποιες ε, αντιφάσεις στην αναφορά. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους άλλους, οι οποίοι δεν είναι ειδικοί για τα οικονομικά ή δεν είναι νομικοί. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε για το επόμενο βήμα. με πιο επακριβή τρόπο οι αναφέροντες να δείξουν ποιοι συγκεκριμένοι νόμοι, κανονισμοί παραβιάζουν τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού πρέπει να συμμορφωθεί η Ουγγαρία, πού πρέπει να προβεί στις δέσσες ε, διορθώσεις. Άρα πιο σαφής διατύπωση. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτή είναι μια θετική πρόταση της συναδέλφου μου, γιατί η Κομισιόν έχει απαντήσει επί τη βάση των πληροφοριών που πρεπει να συμμορφωθει η ουγγαρια που πρεπει να προβει στις δέσμες διορθωσεις διαθέσιμες εκείνη τη στιγμή, ότι δεν υπήρχε κάποια παραβίαση των συνδικών, αλλά τόνισε βάσει των πληροφοριών που είχε εκείνη τη στιγμή σε αυτό το χρονικό σημείο. Αναφέρθηκαν δύο θέματα εδώ πέρα, δύο προβλήματα. Το θέμα της καθυστέρησης των πληρωμών. Εδώ θα ήθελα να ζητήσω από τον αναφερόμενο να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες από την αναφερόμενη καλύτερα για να μπορέσει η Κομισιόν να πάρει μια πιο σαφή θέση για τα θέματα αυτά και μέχρι τότε μπορούμε να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή μέχρι να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Κάτι ακόμα τώρα για, τα, για τις προθεσμίες καταβολής πληρωμών, γιατί έχουμε και άλλη μια αναφορά που θίγει το ίδιο θέμα. Ξέρουμε ότι στον εμπορικό κόσμο μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Κανονικά κάτι το οποίο παραγγέλλεται πληρώνεται, αλλά ξέρουμε πολλές φορές ότι στο δρόμο μεταξύ της παραγγελίας και της ε, πληρωμής μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το ξέρει μερικές φορές κάποιος ότι μπορεί να μην πληρωθεί ποτέ όταν δίδει ένα προϊόν. Στον εθνικό τομέα υπάρχουν δικαστήρια. Εγώ και βλέπω και με ενοχλεί αυτό ότι, και αυτό θα αναφερθεί στην επόμενη αναφορά, πολλές φορές δεν πρόκειται για εμπορευόμενους ή επιχειρηματίες. Πρόκειται για κρατικούς φορείς, για τοπικές αυτοδιοίκησεις οι οποίες καθυστερούν τις πληρωμές τους. Νομίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν θα πρέπει όταν φέρει η αναφερόμενη συγκεκριμένα παραδείγματα ότι στις περιπτώσεις αυτές εάν, να δει στις περιπτώσεις αυτές αν εμπλέκονται και ευρωπαϊκά κονδύλια γιατί εκεί θα πρέπει οι αρχές αυτές να δώσουν και το καλό παράδειγμα δηλαδή εάν έχουν κάνει με ευρωπαϊκά κονδύλια την προκήρυξη της δημόσιας προμήθειας και έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία, θα πρέπει να συμμορφωθούν και με αυτά που λέει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν μπορεί λοιπόν να λένε στους προμηθευτές θα σας δώσω τα μισά και τα άλλα μισά βλέπουμε. Πρέπει λοιπόν να τηρήσουν όλες αυτές οι αρχές τις ε, προδιαγραφές του ευρωπαϊκού δικαίου και θα πρέπει αυτά να τα διευκρινίσει η Επιτροπή να τα διερευνήσει πλήρως και μέχρι τότε να έχουμε πλήρως ότι μέχρι να έχουμε πλήρως αυτά τα στοιχεία να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Πολλές φορές υπάρχει εμπλοκή όχι μοναχα ενό επίπεδου αλλά πολλών επίπεδων διοίκησης και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λεπτομερώς και ενδελεχώς όλα αυτά τα επίπεδα. Κύριος Μποστινάρου, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο μονάχα παρατηρήσεις, πρώτα απ' όλα. Κατά τη δική μου άποψη, και μετά από την πρόταση της Αντιπρόεδρου Χάκης και με την συμφωνία του κυρίου Γιά, θα πρέπει να κατήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Αυτό είναι προφανές. Αλλά προτείνω επίσης να αποστείλουμε και μια επιστολή προς την Ουγγρική κυβέρνηση να μας δώσουν τις δικές τους απόψεις και τη δική τους εκτίμηση για αυτή την κατάσταση και τα μέτρα τα οποία προτείνουν για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Είναι καλύτερα να έχουμε τη θέση της Ουγγρικής κυβέρνησης και τώρα για τα θέματα της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου και του, της μεταγραφής στο εθνικό δίκαιο. Αυτό είναι βέβαια ένα χωριστό θέμα. Αλλά αν μπορούμε να έχουμε μια πλήρη απάντηση από την Ουγγρική κυβέρνηση για τα θέματα αυτά, αυτό θα είναι χρήσιμο όχι μονάχα για τη δική μας Επιτροπή και για την αναφερόμενη, γιατί αυτό θα καταδείξει ότι και η κυβέρνηση της Ουγγαρίας είναι έτοιμη και είναι δεσμευμένη να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα η τελευταία μου παρατήρηση είναι εξής. Θα μπορούσε η Κομισιόν να σκεφτεί τη δυνατότητα να έχει ορισμένες διατάξεις σε σχέση με την προσβασιμότητα των επιχειρήσεων σε, ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκές χορηγήσεις ή σε σχέδια τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχουν κάποιες πιο σαφείς δημοσιονομικές διατάξεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά ούτε οικονομολόγος. Δηλαδή, να μην μπορούν οι δημόσιες αρχές οι οποίες χρωστάνε πάρα πολλά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην μπορούν να έχουν πια πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο μέσα σε μια οικονομική κρίση να βουλιάξει κανεί τι μικρομεσαίε επιχειρήσει από ότι ακολουθώντα αυτή την πρακτική του να μην πληρώνουν τα χρεωστούμενα στι μικρομεσαίε επιχειρήσει δημοσίε αρχέ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Η αναφέρουσα έχει το λόγο για μια πολύ σύντομη απάντηση, σύνοψη. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, πρώτα πρώτα να απαντήσω σε αυτά που είπε η προλαλή Από το 2009 με την προηγούμενη κυβέρνηση υποβάλαμε την αναφορά αυτή. Τότε ήταν τραγική η κατάσταση και μεταξύ 2005 και 2008 είχαμε πάρα πολλές συμβάσεις εις βάρος των ΜΜΕ λόγω των αθεμήτων πρακτικών. Φαντάζομαι ότι παρόμοια και σε άλλες χώρες, αλλά θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό στην ε, Ουγγαρία. Αν θέλουμε να έχουμε καλές συνδικές εργασίες και δίκαιε για τους εργαζομένους, θα πρέπει να εξασφαλίσουν φυσιολογικές συνθήκες εργασίας. Να υπάρχει δίκαιη αμοιβή για εργασία και υπηρεσίες. Αυτό το οποίο εδώ εξηγώ αποσκοπούν στο να τονίσουν κάτι. Ότι πάρα πολλές φορές βλέπουμε το δοκιμάσουν το δίχτυ του σημείου ε σε άλλε χώρε, στο εξωτερικό. Οπότε αυτό μας οδήγησε στη δημιουργία αυτού του δικτύου των εργαζομένων τουλάχιστον πρακτική πολύ κοινή στην ε, χώρα μας. Στο Βέλγιο και, στην Αυστρία βέβαια πάλι υπάρχουν αντίστοιχα μεσάζοντες. Κάτι γνώμη μας αυτοί που θέλουν να βρουν δουλειά φρενάρονται λόγω της, ε, των αδίκων συνδικών αμοιβής εργασίας που επιβάλλουν αυτή η ενδιάμεση. Όλα αυτά τα εξηγούμε στην αναφορά μας. Έχουμε και την αναφορά του 2009 όπου περιγράφεται ότι σας είπα Παρακαλώ, αν κρατήσετε ανοιχτή την αφορά. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε το νομοθέτημα που προβληματίζει. Εάν μια επιχείρηση δεν πληρώνεται από τους ε, χρεώστες της και δεν μπορεί και να προσφύσει τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι πραγματικά ένα πρόβλημα το πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που το μοιράζονται πολλέ χώρε Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ευχαριστώ την αναφέρουσα που παρουσίασε το πρόβλημα αυτό στη συγκεκριμένη επιτροπή. Πιστεύω ότι από τι παρεμβάσει των συναδέλφων μπορείτε να συμπεράνετε ότι υπάρχει μια κοινή θέση όσον αφορά την ανάγκη να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά για να παρακολουθήσουμε και τις περαιτέρω εξελίξεις από πλευρά ιδιωτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω να δέχεστε αυτή την πρόταση να αποσταλεί αίτημα για περαιτέρω πληροφορίες προς τις ουγγρικές αρμόδιες αρχές ελπίζοντας ότι αυτές θα μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία επί των οποίων να βασιστούμε σε πιο συγκεκριμένη αξιολόγηση. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, λοιπόν κλείνουμε τη συζήτηση σε αυτό το θέμα, σε αυτό το σημείο. Ευχαριστούμε την αναφέρουσα. Πάμε στο επόμενο σημείο, την αναφορά του σημείου 10, που είναι η αναφορά 726 του 2010, που υπευλήθη από τον κύριο Ντόχερτη, εξ ονόματι της, ε, των, ε, της Ένωσης Ιρλανδών Οδηγών όσον αφορά το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων στην Ιρλανδία. Είναι παρόν ο αναφέρον, ο κύριος Ντόχερτη, στον οποίο ε, δίνω και το λόγο. My name is John Λέγομαι John Doherty από την Ιρλανδία. Θέλω να σας ευχαριστήσω που δώσατε την δυνατότητα μαζί με τους δύο συναδέλφους μου, συναδέλφους μου να έλθω ενώπιόν σας. Έχουμε στείλει την αναφορά μας και τους τελευταίους έξι μήνες η Κομισιόν δεν μας έχει δώσει κανένα, α, καμία απάντηση και δεν έχουμε ουσιαστικά καμία απάντηση. Νομίζω ότι μας αντιμετωπίζει απαξιωτικά η Κομισιόν για το θέμα του ύψους του τέλους ταξινόμησης και τον τρόπο με τον οποίο καταλογίζονται οι δασμοί στην ε, Ιρλανδία. Εγώ ζήτησα από την Κομισιόν να λειτουργήσει επί τη βάση της αρχής της αναλογικότητας και να σταματήσει αυτή την πρακτική. Ανέφερα μία σειρά από άρθρα της συνθήκης τα οποία πρέπει να τύχουν εφαρμογής για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ έχουμε μία περίπτωση όπου η Ιρλανδία έχει αρνηθεί να εφαρμόσει στοιχεία της συνθήκης ο λαός έτσι χάνει κάθε εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αντίστοιχη πράξη της Ευρωπαϊκής τότε των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 1972 είχαν δώσει μια εξαίρεση στην Ιρλανδία και στη συνέχεια το 1992 η Ιρλανδία απέτυσε το δικαίωμα να δίνει άλλο όνομα σε δασμούς οι οποίοι οδηγούσαν σε απαγορευτική σε απαγορευτικές επιβαρύνσεις αυτούς που θέλουν να εισάγουν αυτοκίνητα στην Ιρλανδία. Ενώ το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλύψει αυτά τα ποσά τα οποία συλλέγει η Ιρλανδία από τους, από τους ειδικούς αυτούς δασμούς. Πού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν γίνεται αυτή η διαδικασία. Υπάρχει κάποια συνωμοσία για να καταλυστευτούν οι πολίτες της Ιρλανδίας από τους δασμούς εισαγωγής. Υπάρχουν 7 διαφορετικές κατηγορίες ε, δασμών που προστίθενται στο ΦΠΑ το οποίο είναι 21% και θα γίνει σύντομα 23%. Αυτό οδηγεί σε τεράστια προβλήματα στην αγορά. Η Mercedes, η Honda, η Seat, έχουν ήδη αποσυρθεί από την αγορά. Αυτό καταδεικνύει ποια είναι η κατάσταση. Όλα αυτά σημαίνουν όμως και μείωση επενδύσεων, μείωση ε, απασχόλησης και δεν επιτρέπουν στους πολίτες Ιρλανδίας να ταξινομήσουν αυτοκίνητα τα οποία θα πιο φιλικά προς το περιβάλλον και πιο ασφαλή και επομένως θα να μειώσουν και τον αριθμό των θανάτων στους δρόμους. Είναι λοιπόν ένας απαγορευτικού χαρακτήρα φόρος ο οποίος επιβάλλεται στα αυτοκίνητα για την ταξινόμηση. Ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο στον Τζέρι. Σας ευχαριστώ. Ίσως να υπάρχει κάποια σύγχυση εδώ πέρα σε σχέση με το φόρο ταξινόμησης και τα τέλη ταξινόμησης. Μπορεί να υπάρχει μια μικρή σύγχυση για τα θέματα αυτά. Οι περισσότεροι στην Ιρλανδία και οι οδηγοί στην Ιρλανδία δεν θα είχαν πρόβλημα αν αγοράζαν ένα αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης να έρθουν στην Ιρλανδία και να πληρώσουν τα κανονικά τέλη ταξινόμησης 100-200 ευρώ όπως εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αγοράζετε το αυτοκίνητό σας για 20.000 ευρώ παραδείγματος χάρη σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και πληρώνετε ένα δασμό 60% πάνω στο ποσό αυτό. πέντε ένα αυτοκίνητο που κάνει 20.000 και πρέπει να πληρώσετε 32.000. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Και οι Ιρλανδοί που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1973 έπρεπε μέσα σε 12 χρόνια να ρυθμιστεί η κατάσταση στην αγορά αυτοκινήτων. Από τότε θα έπρεπε η αγορά αυτή να λειτουργεί από, το από την 1η Ιανουαρίου 1985. Τώρα πλησιάζει η 1η Ιανουαρίου 2012 και δεν είναι ακόμα ελεύθερη αγορά. Πληρώνουμε αυτό το φόρο 36% για την ταξινόμηση αυτοκινήτων. Πιστεύουμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ελέγξει αυτούς τους φόρους που επιβάλλονται και πρέπει να δράσει και να αντιμετωπίσει την κατάσταση που υπάρχει στην Ιρλανδία. Η Κομισιόν δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της και τις υποσχέσεις της και δεν έχει τηρήσει αυτά που αναφέρονται στις συνθήκες γιατί άμα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στην Ιρλανδία, μπορεί να γίνει και σε άλλες χώρες. Έχουμε λοιπόν ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και όχι μόνο ένα Ιρλανδικό πρόβλημα. Okay, excuse me. <clears throat> Now I would like to... Τώρα λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πει κάποια πράγματα. Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είναι μόνο Ιρλανδικό πρόβλημα. Η φορολόγηση των οχημάτων συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν είναι μόνο πρόβλημα της Ιρλανδίας και έχουν υψηλότερου φόρους σε κάποια κράτη-μέλη άλλα. Αλλά το δικαστήριο είπε ότι ευθυγραμμίζεται πλήρω με την νομοθεσία, διότι για την ώρα δεν υπάρχει νόμος Ευρωπαϊκή Ένωσης στον τομέα αυτό, οπότε τα κράτη-μέλη μπορούν να φορολογήσουν σε οποιοδήποτε επίπεδο επιθυμούν από τη στιγμή που δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ αυτοκινήτων που έρχονται από άλλα κράτη-μέλη εν συγκρίση με τα οχήματα που βρίσκονται εντό χώρα. Όπω είπα προηγουμένω, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την περίπτωση. Προσπαθήσαμε με κάποια συνέπεια να αλλάξουμε την κατάσταση. Το 2005 κάναμε πρόταση σχετικά με αυτό, αλλά χρειάζεται ομοφωνία. 27 κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να γίνει αυτό και μέχρι τώρα δεν τα καταφέραμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι για την ώρα δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τις κατασχέσεις, τις κρα... αυτοκινήτων. Ε, δεν έχουμε στοιχεία ότι παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε ερωτήσεις, σχόλια. Κανένας. Ο κύριος Γιάρα, έχετε το λόγο. Ε, Ένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Εδώ βλέπω στη γραπτή απάντηση που αναφέρεται ότι ορισμένες πτυχές του φόρου για την ταξινόμηση είναι αυτή τη στιγμή αντικείμενο μιας διαδικασίας επί παραβάση. Αυτό φαίνεται αντιφατικό. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία, λέει η γραπτή απάντηση, δεν συνάδουν με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν ε, βλέπω λοιπόν πώς μπορούν να συμβαστούν αυτές οι δύο απόψεις. Βλέπω μια αντίφαση. Εγώ φαντάζομαι ότι είναι πράγματι κάτι το οποίο θίγει τα συμφέροντα των καταναλωτών όταν υπάρχει ένας τέτοιος φόρος του ύψους του 36%. Μπορεί να επιμείνουν κάποιοι να πούν ότι οι Ιρλανδοί ήταν πιο έξυπνοι, καταφέραν να έχουν μια μεταβατική περίοδο, αλλά σε τελική, ε, σε τελική ανάλυση ο δασμός εισαγωγής έχει αντικατασταθεί από ένα φόρο ταξινόμησης. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αξιοπρεπές από την πλευρά μιας κυβέρνησης. Αυτό πρέπει να πω. Αλλά θα ήθελα να υπάρξει και μια διευκρίνηση αυτής της αντίφασης που λέτε εσείς ότι δεν υπάρχει παραβίαση συνθήκη, ενώ η, η γραπτή απάντηση λέει ότι πράγματι υπάρχουν κάποια τέτοια στοιχεία. Αυτή είναι η 0726. Η αναφορά αυτή δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι η γραπτή απάντηση αναφέρει ότι υπάρχει κάποια... Η τελευταία στήλη, η τελευταία γραμμή μάλλον, οι ε, τελευταίες γραμμές αναφέρουν ότι υπάρχουν στοιχεία παραβίαση των συνδικών. Άλλα ερωτήματα, άλλα σχόλια. Η... Αν δεν έχετε άλλα σχόλια, θα ζητήσουμε από τον αναφέροντα να μας πει αν έχει κάποια σχόλια. Yes, I would like to reply to that there. Να απαντήσω. Στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής if realizes what... Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει η αρχή της αναλογικότητας. Με κατάσχεση αυτοκινήτου που κοστίζει 20.000 για 5.000 δεν μπορείς τελικά να, να, να, να βρεις την αντιστοιχεία. Μόνο το αντίστοιχο μπορείς να πάρεις. Δεν μπορείς για ένα αυγό να πάρεις μια ολοκληρικότητα. Χρειάζεται αναλογικότητα. Αυτό εννοούμε. και παρεκκλήσεις τώρα εξαιρέσεις. Έχουμε δεκαετή παρέκκληση πήραμε όταν πρωτομπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώδεκα χρόνια αργότερα έπρεπε να εκπνεύσει. Ε, συνεχίστηκε και άλλαξε τον όρο των τελωνιακών ε, δασμών. Πρέπει να διαβάσει κανείς τους όρους της συνθήκης. Στα άρθρο 25 αναφέρεται ότι τελωνιακή δασμοί θα απαγορεύονται και οι συναφείς φόροι και αναδιαπο... αναδιατύπωσαν τον τελωνιακό δεσμό και επιβάλλουν τον ίδιο φόρο. Λοιπόν, με άλλη ονομασία εισπράττονται τα ίδια τέλη. και επέβαλαν αντίστοιχο ε, ΦΠΑ τελικά, τόσο ώστε να αντισταθμίσουν τον καταργηθέντα φόρο. Αυτό έχει συνέβη. Ευχαριστώ. Το δεύτερο τμήμα. Σημείο 11. Η αναφορά αυτή είναι παρόμοια. Είναι σαν το δεύτερο μέρος του ιδίου ζητήματος. Um Θέλω και πάλι να παρακαλέσω την Κομισιόν να διευκρινίσει. Είπε σήμερα η Κομισιόν ότι όλα αυτά συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η γραπτή απάντησή της λέει κάτι διαφορετικό. Παρακαλώ να, να διαλύσει αυτή την παρεξήγηση, αν παρεξήγηση, ή να διευκρινίσει αυτή τη φαινομενική αντίφαση. Γιατί αναφέρεται ότι στην γραπτή απάντηση ότι τμήματα αυτή τη ε, προβληματική αποτελούν στοιχεία μια διαδικασία επί παραβάση. Είναι αλήθεια ή όχι. Παρακαλώ να μου εξηγήσει η Κομισιόν γιατί η προφορική του απάντηση είναι διαφορετική από τη γραπτή του απάντηση. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Μπλουμ από την Κομισιόν να απαντήσει. Δεν υπάρχει εναρμόνιση. Δεν υπάρχει επομένω θέμα εφαρμογή του ευρωπαϊκού κοινωνικό δικαίωμα να κάνουν όμως ό,τι θέλουν τα κράτη-μέλη. Ό,τι φορά θέλουν, επιβάλλουν, αρκεί να υπάρχει δεσμενής διάκριση. Επίσης κρίνει το δικαστήριο ότι αυτό δεν είναι δασμός τελωνιακός τέτοιου είδου ε, τέλος. τώρα το άρθρο 113 όσον αφορά τα θέματα της παραβιάσεως του κοινωνικού δικαίου Το θέμα είναι αν κανεί ε, νοικιάσει ένα αυτοκίνητο κάπου αλλού και θα το χρησιμοποιήσει στην ε, Ιρλανδία, τότε, τότε έχουμε διαδικασία παραδάση. Και επίση έχουμε και απομείωση αξία των ε, νεωτέρων από τριών μηνών αυτοκινήτων. Ναι, ευχαριστούμε και τώρα έχουμε το, άλλο θέμα. Μπορείτε να απαντήσετε. Α, όχι. Έχουμε τίποτα άλλο, όχι επομένως. No, this issue. I μπορεί να to αυτό. All members wish to close it at this stage. No, I, I asked, but open. keep open. The petition keep open. Yes. Hold... Θα παραμείνει λοιπόν ανοιχτή η αναφορά. Η συζήτηση σταματά, αλλά παραμένει ανοιχτή η αναφορά. Yes. Yes, I would like to ask Mr. Stewart. Ο κύριος Stewart έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε, σας πειράζει να ακουστούν και οι δύο αναφορές ταυτόχρονα. Μιλάω εκ μέρους του Πολ Μακόλγκαν και για τον εαυτό μου όσον αφορά τις δύο αυτές αναφορές. Είμαστε, ζούμε κοντά στα σύνορα, είναι παραμεθόρια περιοχή εκεί που ζούμε. Δύο νομοθεσίες αναμειγνύονται λόγω απασχόλησης, λόγω οικογενειακής ζωής, λόγω κοινωνικών πτυχών και στις συνοριακές περιοχές, παραμεθόριες περιοχές, τι αντιμετωπίζουμε. Διαφορετικές νομοθεσίες που αλληλεπικαλύπτονται. Όσον αφορά τον κύριο Μακόλγκαν, ε, εργάζεται στη Βόρεια Ιρλανδία, κάνει, ασχολείται με διάφορες απώλειες και αποζημιώσεις και πρέπει να έχει όχημα καταγραμμένο ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχει πρόβλημα να πληρώνει το τέλος ταξινόμησης, έχει και άλλα δύο οχήματα που είναι καταχωρημένα στην Ιρλανδία. Αλλά για τη δουλειά του Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα όχημα που είναι καταχωρημένο στη Βόρεια Ιρλανδία. Του δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Παραβιάζει τον νόμο σε αυτή τη φάση. Στη δημοκρατία για να πάει στη δουλειά του. Αν ήθελε να οδηγήσει το όχημά του που είναι καταχωρημένο στη Νότια Ιρλανδία θα υπόκειτο σε πειθαρχική δράση και πιθανώ σε απόλυση. Το να λέμε ότι είναι απλώ ασφαλιστικό θέμα αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όταν μάλιστα ο κύριος έχει πληρώσει φόρο ταξινόμησης δύο φορές σε δύο διαφορετικά οχήματα. Το να διατείνεται κανείς ότι υπάρχει παραβίαση των όρων απασχόλησής του ε, είναι κάτι πολύ τραβηγμένο. Ζούμε τόσο κοντά στα σύνορα, βλέπετε. Και βλέπουμε διαφημίσεις, αγγελίες ιστοσελίδες και σε εφημερίδες όπου εταιρείε στη Βόρεια Ιρλανδία διαφημίζουν να βρουν κόσμο που θα πρέπει να έχει το δικό του αυτοκίνητο. Διότι πρέπει να έχουν καταχωρημένα οχήματα στη Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε οι Ιρλανδοί τι Δημοκρατία τη Ιρλανδία δεν μπορούν να πάρουν αυτέ τι θέσει. Αν είναι θέμα συνοριακή απασχόληση, θα έπρεπε να υπάρχει παρέκκληση από την Ιρλανδική κυβέρνηση, τους, ώστε ο κόσμο να μπορεί να συμμετέχει. Έχουμε, είναι περιοχή 15% ανεργία. Αν θέλουν κάποιοι να φύγουν από την ανεργία και να δουλέψουν και να πάνε σε γειτονική χώρα, εγώ νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ λογικό. Τώρα στη δική μου αναφορά πάω. Ήρθε σε επαφή μας. Ήρθε σε επαφή εκατοντάδες φοιτητές μαζί μου. Ξανά μιλώ για παραμεθόρια περιοχή. Έχουμε ντόπιου φοιτητέ που πάνε στο Belfast για πανεπιστήμιο, για σπουδές και επειδή οι υπεύθυνοι εισοδήματο της Ιρλανδίας θεωρούν ότι ο τόπος διαμονής είναι ο, ο τόπος κατοικίας τους δεν μπορούν να οδηγήσουν σε δύο δικαιοδοσίες ταυτόχρονα. Η ασφαλιστική εταιρεία παίρνει τη διεύθυνση διαμονή του Πανεπιστημίου σαν τόπο διαμονή κανονικό, ενώ υπεύθυνοι του Υπουργείου Οικονομικών τον τόπο της, το σπίτι του, το οικογενειακό. Αν ένα Ιρλανδό πάει στο Μπέλφαστ με το όχημά του καταχωρημένο στη Δημοκρατία τη Ιρλανδία, επειδή το έχει στα χέρια του για, γιατί μένει στο Μπέλφα στη Βόρεια Ιρλανδία για πάνω από 185 μέρες δεν έχει σωστή ασφάλιση. Απ' την άλλη, αν οδηγήσουν όχημα με πινακίδες βόρεια Ιρλανδίας που θα πρέπει να, να κάνει τεχνικό έλεγχο στο Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνει ασφάλιστρα Ηνωμένου Βασιλείου ε, τέλη κυκλοφορία Ηνωμένου Βασιλείου. Αν πάει το στο σπίτι του, τότε θα του το κατάσχουν οι Ιρλανδοί ε, το όχημά του, γιατί δεν έχει πληρώσει το τέλο ταξινόμηση. Άρα στην περίπτωση ταινία κάτσε 22. Δεν έχουν σε αδιέξοδο, δεν έχουν λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι οι ξένοι σπουδαστέ που πάνε στη ε, Δημοκρατία τη Ιρλανδία εξαιρούνται, θα πρέπει να υπάρχει και το αμφίδρομο, το αντίστροφο. Και οι Ιρλανδοί και διασυνοριακοί εργαζόμενοι που διαμένουν κατά διάρκεια της εβδομάδας ε, μακριά από το σπίτι του θα πρέπει να ωφελούνται από μια εξαίρεση από αυτόν τον νόμο. Σε πρώτερη υπόθεση που εξετάστηκε από την Επιτροπή η οδηγία 83-182 ΕΟΚ στο άρθρο 7 7-1 της οδηγίας λέει ποιος είναι ο τόπος διαμονής. Εκεί που συνήθως μένει κάπως και τουλάχιστον 185 μέρες ε, σε κάθε ημερολογικό έτος. Αυτό είναι συνηθιστό όπως κατοικία. Άρα είναι αντίθετο με αυτό που κάνει η Δημοκρατία της Ιρλανδίας που λέει στους φοιτητές. Ε, το καταλαβαίνω αν Ιρλανδοί φοιτητέ έχουν κάποια υποτροφία που χορηγείται από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Αν δεν υπάρχει όμως άλλος δεσμός, δεν μπορεί να διατείνεται η δημοκρατία της Ιλλανδίας παρόλο που περνάει τα δύο τρίτα του έτους σε άλλη α, χώρα μέλος ότι σύνδεσμος τόπος διαμονής είναι η δημοκρατία της Ιλλανδίας. Και λέει, να επανέλθω στο κείμενο, το άρθρο 7.1 της οδηγίας θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι εννοεί ότι όποιος έχει προσωπικούς και ε, εργασιακούς δεσμούς με ένα κάτω μέλος είναι σύνδεσμος τόπος διαμονής. και τα το κέντρο μονίμων συμφερόντων που βρίσκονται. Γίνεται αξιολόγηση. Πρέπει να εντοπιστούν που ήταν τα βασικά του συμφέροντα. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να καταλήξουν κάπου, πρέπει να, το, να σταθμιστούν οι προσωπικοί δεσμοί. Μπορεί να είναι κάποιο φοιτητή, ο οποίο να φεύγει από την Ιρλανδία για μόνιμα. Άρα, ουσιαστικά δεν έχουν δικαίωμα με την κατάσταση άλλο κάτω μέλο οι Ιρλανδοί τη Δημοκρατία Ιρλανδία. Δηλαδή, οι προσωπικοί δεσμοί εκεί επικρατούν. Παρόλο που στα άρθρο 7.1 λέει ότι είναι για 185 μέρε. Τα χρησιμοποιούν και ασφαλιστικέ εταιρείε αυτά τα κριτήρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι είπε. Ότι η εξαίρεση θα οδηγούσε στο να θα γινόταν κυνήγι ε, με το χαμηλότερο επίπεδο φορολόγηση. Θα πήγαιναν όλοι να καταχωρήσουν τα οχήματά του στη χώρα που έχει χαμηλότερη φορολόγηση. Από την άλλη πλευρά, αν τα ασφάλιστα σε μια χώρα είναι πολύ χαμηλότερα από άλλα κράτη-μέλη, Μπορεί ένα άτομο, α πάρουμε τη Γαλλία, αν η Γαλλία είχε το χαμηλότερο ασφάλιστρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σταματά τον Ιρλανδό να πάει εκεί να ασφαλιστεί. Το ότι ασφαλιστική δεν θα δεσμευτεί διότι υπάρχει κίνδυνος που συνεπάγεται, ξεπερνάει τις 185 μέρες που δεν διαμένει στη χώρα ο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έκτοτε έλαβα και άλλες πληροφορίες του Υπουργείου Οικονομικών της Ιρλανδίας. Αυτά που λένε υποστηρίζουν αυτά που λέω. Είναι φραγμός αυτό για το ελεύθερο εμπόριο. Να σας διαβάσω και την απάντηση, ένα κομμάτι της απάντησης. 18 μήνες πολεμώ για το θέμα αυτό στην Ιρλανδία. Και λέει επιστολή. Περιέγραφα πώ θα ήταν υποφελέ για τα αυτοκινητομηχανία στην Ιρλανδία αν υπήρχε απαλλαγή από το τέλο ταξινόμηση. Και ποια απάντηση μου δόθηκε. πλησιάζει στην παραδοχή ότι χρησιμοποιούν αυτό το τέλος σαν ένα εμπόδιο στο ελεύθερο εμπόριο. Η παράγραφος έχει ως εξή. Η κατάργηση του VRT δεν θα φέρει σε καλύτερη θέση τους εμπόρους αυτοκινήτων μέσω και μακροπρόθεσμα. Ίσως να είναι φθηνό το αυτοκίνητα πριν το φόρο, αλλά ίσως λόγω όγκου ε, πωλήσεων το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορεί να ανταγωνιστεί καλύτερα στην ελληνική αγορά, οπότε θα κάνει πιο μακροπρόθεσμη ζημιά στην αυτοκινητοβιομηχανία τη βιομηχανία στην ε, Τη Ιρλανδία, παρόλο που θα μπορούν να προσφέρουν καλύτερα αυτοκίνητα σε καλύτερε τιμέ οι, οι πολιτές του Ηνωμένου Βασιλείου από ό,τι οι Ιρλανδοί. Αν αυτό δεν είναι παραδοχή δεν ξέρω ποιο πράγμα είναι παραδοχή ότι αυτό είναι φραγμός στο ελεύθερο εμπόριο. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. για την παρουσίασή σας, η οποία ήταν σαφέστατη νομίζω. Κυρία Βρούμ, έχει το λόγο από την Κομισιόν. Και πάλι. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Κομισιόν θέλει πράγματι να βρει μια λύση για να αποφύγουμε μια τέτοια κατάσταση χωρί εναρμόνιση. Αλλά μέχρι στιγμή έχει καταστεί αδύνατο γιατί τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν. Για την πρώτη αναφορά, είπε το δικαστήριο ότι δεν χρειάζεται να ταξινομείτε ένα εταιρικό αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν χρειάζεται να, να ταξινομηθεί αλλού αν το χρησιμοποιείτε σε ένα κράτος μόνιμα. Σε αυτή την περίπτωση όμως όταν πρόκειται για ιδιωτικό αυτοκίνητο τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν ένα φόρο ταξινόμησης εφόσον δεν έχει διακριτικό χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια αυτοκινήτων υπάρχει η συμβατική ελευθερία των ασφαλιστικών εταιρείων και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα η Κομισιόν για την διστακτικότητά τους να ασφαλίζουν αυτοκίνητα κάτω από ορισμένε συνθήκες. Για τη δεύτερη αναφορά, την 1357, θα έλεγα ότι όταν ένας φοιτητής χρησιμοποιεί ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο που είναι ταξινομημένο στην, ε, στο φυσιολογικό τρόπο διαμονής του και το χρησιμοποιεί σε ένα άλλο, άλλο κράτος όπου σπουδάζει, έλκεται από το άρθρο 5 της οδηγίας που ανάφερε ο αναφερόμενος ότι το αυτοκίνητο αυτό δεν θα πρέπει να πληρώνει επιπλέον φόρο ταξινόμησης. Και εδώ η Ιρλανδική νομοθεσία είναι ευθυγραμμισμένη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Απλώς φαίνεται ότι οι Ιρλανδικές εταιρείες ασφάλισης δεν θέλουν να ασφαλίσουν το αυτοκίνητο και έχουν πράγματι την ελευθερία συμβατικής, συμβα, τη συμβατική ελευθερία και δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπλουμ, παρακαλώ. Κύριε Μπουστινάρου. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο δύο λόγια για άλλη μια φορά. Φοβάμαι ότι εδώ πέρα βασιλεύει σύγχυση. Για να σας τα πω στα ρουμανικά, γιατί υπάρχουν κάποιοι τεχνικοί όροι που καλύτερα θα σας τους πω στην γλώσσα μου. Πρώτα πρώτα. Πρώτα πρώτα θέλω να σας πω ότι είναι παράδοξο το ότι αυτή η πράσινη κάρτα που επιτρέπει στα αυτοκίνητα με διεθνή ασφάλιση να πάνε σε άλλη χώρα δεν δουλεύουν στα σύνορα Βορείου Ιρλανδίας και Δημοκρατίας Ιρλανδίας. Αυτό θα πρέπει όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε εδώ πέρα άσκηση μονοπωλίου από ασφαλιστικές εταιρείε γιατί αρνούνται να ασφαλίσουν αυτοκίνητο σε ένα άλλο χώρο. Αυτό επομένως οδηγεί σε αύξηση των ε, εξόδων για τους οδηγούς. Δεν θέλω να μιλήσω σαν πολιτικός. Πάντως θεωρώ ότι το να γίνονται τέτοια πράγματα αυτό είναι φραγμό στην ελευθερία διακίνηση ε, προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη δεν είναι μόνο για ελεύθερη κυκλοφορία. Για μια αρχή ελεύθερη κυκλοφορία λέει για ένα δικαίωμα το οποίο θα πρέπει να ασκείται χωρί κανένα φραγμό και να το απολαύουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Άμα εγώ σα λέω ότι δεν μπορείτε να περάσετε την άλλη πλευρά των συνόρων για να δουλέψετε, αν δεν έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο να έχει πινακίδε όπω εγώ ορίζω και να είναι και ασφαλισμένο όπω εγώ θέλω, όπω θέλει το καθένα. Ε, αυτό είναι σαφώ ένα φραγμό στην ελευθερία τη κυκλοφορία όπω την ορίζει η συνθήκη. Τρίτον, Εδώ πέρα έχουμε δεσμενή διάκριση από πλευρά του εργοδότου σε σχέση με κάποιον δυνάμει εργαζόμενο. Διότι τάσσονται εδώ κάποιε ε, προποθέσει σε σχέση με την ε, νόμιμη κατοικία και τι πινακίδε του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί ο για να πάει στη δουλειά του. Και αυτό αφορά του όρου προποθέσει που όσον αφορά την ε, ασφάλιση του αυτοκίνητου που για να πάει δουλειά. Εμεί εδώ πέρα πρόκειται για τριπλή τη μενή διάκριση και άλλο αυτό πρέπει να το εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να επιληφθεί αυτό, θα πρέπει να κάνει τι αναγκαίε ενέργειε. Αυτό είναι καυκικό. Καλύτερο στον Νέο Κάφκα θα περιγράφει από αυτά τα οποία γίνονται τώρα το 2011 και μεταξύ Αγγλίας και Ιρλανδίας. Είναι δυνατόν τα σύνορα εκεί να δημιουργούν τέτοιο πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα να κινδυνεύει να επιθέσει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι, είναι παράλογο. Και επίση αποτελεί ένα πρόβλημα για την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων. Ωραία όλα αυτά που είπαμε τώρα. Όμω, έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανέκαθεν ναι, ε, λέμε ότι ένα φόρο θα πρέπει να είναι εύλογο. Δηλαδή να είναι δυνατόν να καταβληθεί από τον πολίτη, από τον φορολογούμενο, αυτό τον οποίο υποχρεωτεί να το καταβάλει. Επομένω, ο φόρο θα πρέπει επίση να είναι αναλογικό σε σχέση με τι ε, υπηρεσίε που προσφέρονται στη συνέχεια χρησιμοποιώντα το φόρο πλευρά του κράτου. Δηλαδή, δεν είναι αυτό η προσωπική μου ανακάλυψη. Από την Γαλλική Επανάσταση έχουμε αυτή την ε, αρχή και τη χρησιμοποιούμε συνέχεια. Έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή και μα λέει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να προβαίνουν σε τέτοιου είδου ε, παράλογες ε, ε, φορολογήσεις. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει ούτω ώστε και για τους φόρους να ισχύει το εύλογο και η αναλογικότητα. Και αυτό ισχύει για όλους, για τους Ρωμάνους, τους Ιρλανδούς. Να μπορεί δηλαδή κάποιος να έχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Γι' αυτό το λέμε και ενιαία αγορά. Μα είναι δυνατόν να έχουμε ένα φόρο ο οποίο να ανέρχεται στο 60% τη ε, αξία πωλήσεω ενό προϊόντο. Εν προκειμένου μιλάμε για την αξία, την τιμή του αυτοκινήτου. Εδώ έχουμε κατάφορη παραβίαση τη κοινωνική νομοθεσία, οπότε σα παρακαλώ και εσεί Κομισιόν και εμεί εδώ θα πρέπει να βγούμε αυτή την κατάσταση. Κυρία Πρόεδρε, τα ξέρετε καλά. Βεβαίως και να επενετεί η Κομισιόν. Μάλιστα είχε κάνει και εκείνο το τελεσίγραφο προς τη Ρουμανία όσον αφορά το τέλος κυκλοφορίας, το οποίο ήταν ε, ε, αντίθετο στο κινητικό δίκαιο, στη Οπότε συνεντουσιάστηκαν οι Ρουμάνοι και είπαν να, να, που σε κάτι χρησιμοποιεί η Ευρώπη, σε κάτι συγκεκριμένο. Όμως εν προκειμένου ερχόμαστε και λέμε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί τίποτα να κάνει. Θεατισμένη στι ενέργειες ενός ε, κράτους το οποίο επιβάλλει τέτοιου τερατώδης τερατώδει εις τους πολίτες του. Αφόρητος αυτός ο φόρος για του περισσότερου Ιρλανδούς. Προλογμένως επόμενος το πέρα είναι το θέμα. Είναι να κάτσει κανείς και να κατανοήσει τι θέλει να πει η συνθήκη και τι θα είναι το κοινωνικό δίκαιο. Ε, thank you. Ε, Εμεί σα ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Oh, excuse me, please. Äh, Πάρα πολύ σύντομα. Μπερδεύουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η φορολογία και το άλλο είναι η ασφάλιση των αυτοκίνητων. Δεν πρέπει να τα συγχαίρουμε και τα δύο. Γιατί αυτό θα οδηγήσει σε μία σύγχυση. Και δεν ξέρω αν έχω καταλάβει πλήρως την κατάσταση που επικρατεί. Προφανώς εδώ εμπλέκονται θέματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την ενιαία αγορά και με την ελεύθερη κυκλοφορία. Δηλαδή υπάρχουν ρυθμίσεις που δεν έχουν καμιά σχέση με αυτές τις αρχές. Γι' αυτό προτείνω να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και ίσως θα ήταν χρήσιμο να πάρουμε και κάποιες πιο εμπεριστατημένες πληροφορίες από την Επιτροπή μεταφορών και ενδεχομένως να μας δώσουν και κάποιες προτάσεις. Αν πρέπει κανείς όταν μένει σε ένα άλλο κράτος μέλος να πρέπει να πληρώνει, ε, να πληρώνει επιπλέον φόρο, ταξινόμηση και όλα αυτά, όλα αυτά φαίνονται πάρα πολύ μπερδεμένα. Ήθελα λοιπόν να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την ε, οδηγία και να ζητήσουμε από την αρμόδια επί της επιτροπή, την Επιτροπή Μεταφορών, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και μετά να έρθουμε σε συζήτηση πάλι με την Κομισιόν. Δεν θέλω αυτό το θέμα να μπει στο αρχείο. Αυτό δεν θα βοηθήσει κανένα. Πρέπει να μας απασχολήσει και να μας βοηθήσει και η Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ. Κύριε Γιά, νομίζω και εγώ ότι πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και μια πρόταση αντίστοιχη με αυτό που αναφέρατε είναι ότι πρέπει να στείλουμε και μια επιστολή στις, ε, Αγγλικές, στις ε, Ηνωμενοβασιλιώτικες και τις ελληνικές αρχές να ζητήσουμε επίσης και την ε, άποψη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Επόμενο θέμα είναι το σημείο 12 του Λόρδου Richard Inglewood για το, τη διάκριση που εισάγει ο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2008 για την έκπτωση από το αξίωμα του μέλους της βολή των Λόρδων, μελών που έχουν εκλεγεί βουλευτές του ΕΚ. Παρακαλώ. Ο κύριος Τσίτσεστερ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αναφορά αυτή προέρχεται από ένα πρώην συνάδελφο, τον Λόρδο Ίγκλεγουτ. Μπορεί να σας φαίνεται αυτό ότι είναι ένα θέμα ε, κατά κάποιο τρόπο αποκρυφιστικού χαρακτήρα. Αλλά υπάρχει μια, μεγάλη, μια σημαντική αρχή η οποία εμπλέκεται εδώ, ότι τα μέλη της Βουλής των Λόρδων που έχουν το χαρακτήρα ισόβιου μέλους της Βουλής των Λόρδων δεν μπορούν να έχουν μια εξαίρεση εάν θέλουν να είναι υποψήφοι για εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή κάπου αλλού. Τα αντίθετα, τα κληρονομικού χαρακτήρα μέλη της Βουλής, της Βουλής των Λόρδων δεν έχουν μια τέτοια εξαίρεση. Και ο Λόρδος Σίγκλεγουτ θεωρεί ότι αυτό αποτελεί μια διάκριση βάσει του άρθρου 20, ρήτρα 2β, άρθρο 2β, των συνθήκων αναφέρεται στη σελίδα 83, 5, 6 λέει ότι έχει ως δικαίωμα ο Ευρωπαίος πολίτης να είναι υποψήφιος για εκλογή σε ένα άλλο κράτος μέλος και να εκλεγεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν γίνει αυτό βάσει των εθνικών διατάξεων. Αλλά βάσει των διατάξεων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος σε άλλο κράτος μέλος και λέει ότι αυτό είναι μια διάκριση γιατί αφορά μονάχα ένα τμήμα των μελών της Βουλής των Λόρδων. Από ό,τι κατανοώ τώρα από τα σχόλια της Κομισιόν τους ανέφεραν οι Βρετανικές αρχές ότι το θέμα αυτό καλύπτεται από ένα σχέδιο νομοθεσίας για την μεταρρύθμιση της Βουλής των Λόρδων που είναι υπό εξέταση στο Ηνωμένο και αυτό μπορεί να είναι ε, μια δικαιολογία για να μην κάνει κανείς τίποτα και να αφήσει το πρόβλημα να λυθεί από μόνο του. Αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η μεταρρύθμιση της Βουλής των Λόρδων στο Ηνωμένο Βασιλείο είναι μια διαδικασία που κρατάει πάρα πολύ χρόνο. Ξεκίνησε πριν από καμιά εκατονταετία περίπου και μπορεί να κρατήσει άλλη με άλλο ένα αιώνα. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο πολιτικό θέμα και εμπλέκονται πολλά πολιτικά συμφέροντα. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι τουλάχιστον κυρία Πρόεδρε θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και να ελέγξουμε πράγματι κατά πόσον οι Βρετανικές αρχές θα προχωρήσουν σε μια μεταρρύθμιση των κανόνων που διέπουν τη Βουλή των Λόρδων ή ακόμα και να τους πιέσουμε να προχωρήσουν σε μεταρρύθμιση σε σχέση με το συγκεκριμένο αυτό σημείο. Γιατί το γενικό θέμα της μεταρρύθμισης της Βουλής των Λόρδων θα χρειαστεί πολύ χρόνο να κατασταλάξει και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο Λόρδος Ιγκλεγουτ δεν θα έχει την δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του εν ευθέτω χρόνο. Αν θέλετε άλλες λεπτομέρειες είμαι στη διάθεσή σας. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Κομισιόν για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Όκεν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μ' αρέσει αυτή η αναφορά, μ' αρέσει να την κρατάω ανοιχτή. Ε, μ' αρέσει. Επίσης ότι κανονικά δεν νομίζω ότι έπρεπε να παρεμβαίνουμε στην νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό πιστεύω. Αν έχει νόμους το Ηνωμένο Βασίλειο που σας δημιουργούν προβλήματα και νομίζω ότι κάτι δεν συμβαίνει. Ε, μόνο από το Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται η αλλαγή. Δεν έχετε καν σύνταγμα. Και ακούγεται σαν θέμα που αφορά συνταγματική αλλαγή. Ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν δημιούργησε ο Θεός το σύστημα και θα μπορούσε να αλλάχθεί από τους πολίτες αυτή τη ε, δημοκρατία που είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχω σοβαρό πρόβλημα παραμείνει ανοιχτή. Ε, μ' αρέσει. Θα με έθλιβε τα μάλα αν έκλεινε αυτή η αναφορά. Κύριο Μποστινάρου, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινώντας από αυτό που είπε η αγαπητή συνάδελφος, η κυρία Άουκεν, ας κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή μέχρι ότου η Βουλή των Λόρδων να βρει νομική λύση για το πρόβλημα. Θα είναι εξαιρετικό αυτό ως λύση για όλους τους ευρωβελευτές. Σε 200 χρόνια ίσως έχουμε απάντηση. Αλλά τώρα ας μην αστευόμαστε. Κι άλλο συμπέρασμα υπάρχει. Πάρα πολλά opt-out είναι εις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών μας που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αλλού. Απευθύνω έκκληση. Οι ευρωπαϊκοί νόμοι και οι κανονισμοί να εφαρμόζονται πανταχού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι υπέρ του να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Σοβαρά τώρα. Διότι εδώ παραβιάζεται ένα δικαίωμα που ανήκει σε άτομα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. κύριος Γιάρ. Ε, ε, να προσθέσω και το εξή. Να την κρατήσουμε ανοιχτή, αλλά όχι για 200 χρόνια. Θα πρέπει όλοι μαζί να δούμε, να λύνεται αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, να την κρατήσουμε ανοιχτή, αλλά όχι στο σε αυτή την αναφορά, επομένω. Ο κύριος Τσίτσεστερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μόνο να προσθέσω το εξής. Εδώ τίθεται θέμα του να ενθαρρύνετε, να παροτρύνετε τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να κάνουν κάτι, κάτι το οποίο το έχουν κάνει ήδη σε σχέση με τους ισόβιους λόρδους. Αυτό επέτρεψε στην συνάδελφό μας την Λέδη Λάτφορντ να παραμείνει μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και έχει τη δυνατότητα όταν τελειώσει η θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξαναγυρίσει στην Βουλή των Λόρδων. Υπήρξε λοιπόν σε μια προηγούμενη κυβέρνηση μια τέτοια ρύθμιση. Ελπίζω ότι τώρα η τωρινή κυβέρνηση θα αποφασίσει να άρει αυτή την ειδική κατάσταση που υπέδειξε ο Λόρδος Σίγκλεγουτ. Είναι θέμα αρχής λοιπόν και ελπίζω ότι πρώτα θα κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και δεύτερον θα μπορούσαμε να ζητήσουμε πληροφορίες από τις Βρετανικές Αρχές για το πόσο χρόνο θα χρειαστούν για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ωραίο γράμμα το οποίο θα μπορούσατε να αποστείλετε εσείς κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ να το δω. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία που υποστηρίζει το να παραμείνει ανοιχτή εν λόγω αναφορά. Την αφήνουμε ανοιχτή την αναφορά. Και θα υποστηρίξω και το αίτημα του συναδέλφου του κ. Τσίτσεστερ να αποσταλεί και άλλο ένα σημείωμα προς διευκρίνηση προς τις Βρετανικές Αρχές να μας διευκρινίσουν τουλάχιστον πόσο καιρό πρέπει να περιμένουμε για να αλλάξει νομοθεσία. Αν δεν θέλει άλλος να παρέμβει, μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση επί της τελευταίας αναφοράς και κάνα δεκάλεπτο θα διακόψουμε περιμένοντας να πάει 5.30 για να ξεκινήσει η συνέδριση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ όλους.